Bonjour, chers collègues. Nous Καλημέρα σα, συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με το 7 τη ημερήσια διάταξη. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για τη μεταφορά προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του ειδικού δικαστηρίου για τους ε, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε δημιουργηθεί. Γενικά δεν θα κάνουμε τη συζήτηση από την αρχή, η συζήτηση έγινε πέρυσι, αλλά η πρόταση αυτή στην ουσία περιλαμβάνει τις ιδέες οι οποίες ε, είχαν εκφραστεί σχετικά με την απορρόφηση των επτά δικαστών του δικαστηρίου αυτού στο ευρύτερο παλαιότερο δικαστήριο από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016. Πρόκειται δηλαδή ε, για μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Προτείνουμε κάποιες τεχνικές, τεχνικού τύπου τροπολογίες σχετικά με τη νομική βάση επί της οποίας λαμβάνεται η απόφαση. Η δική μας νομική υπηρεσία θεωρεί ότι η νομική βάση την οποία προτείνει το δικαστήριο δεν είναι η σωστή. Γι' αυτό γίνονται κάποιες αυστηρά τεχνικές τροπολογίες που δεν αφορούν στο περιεχόμενο ε, της ρύθμισης. Στην έκθεσή μας κάνουμε ορισμένες συστάσεις σχετικά με την μεταβατική περίοδο, γιατί όπως είπα από την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υπάρξουν οι μεταφορές των δικαστών. Συστήνουμε επίσης προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αναδιοργανώσει τις εργασίες της από την 1η Σεπτεμβρίου. Θα είναι ένα δικαστήριο με 47 δικαστές, οπότε μπορεί ε, να έχει περισσότερα δικαστήρια ανοιχτά με πέντε δικαστές το καθένα, έτσι ώστε να δοθεί ένας ε, ρυθμός ε, καλύτερος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν θα υπάρχει λοιπόν ειδικό δικαστήριο, αλλά μπορεί ένα τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να συγκεντρώνει τα θέματα ανάλογα με, το, με την ύλη, με την φύση Κάτι το οποίο θα επιτρέψει σε, μια συγκεκριμένη, σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δικαστηρίου να αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη και να αυξήσει την ταχύτητα με την οποία λαμβάνει τις αποφάσεις του. Αυτά είναι. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, άλλα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συζητήσουμε. Η προθεσμία είναι η 23η Μαρτίου για την κατάθεση των τροπολογιών. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά λέει και ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κυρία Ντελβό. Ο κύριος Ζήφκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντελβό για την εξαιρετική της προσπάθεια. Έχουμε να διανύσουμε το τελευταίο αν θέλετε βήμα, να κάνουμε μάλλον το τελευταίο βήμα για την αλλαγή αυτή. Συμφωνώ με τις συστάσεις της εισηγήτριας, πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η έκθεση αυτή είναι τεχνικής φύσεως και δεν χρειάζεται εδώ να ξεκινήσουμε σχόλια στις προτάσεις της εισηγήτριας. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω κατά κάποιο τρόπο με, σε πολιτικό επίπεδο για την πρόταση αυτή. Εγώ στην έκθεση αυτή θα ήθελα να υπάρχουν ορισμένα επιπλέον στοιχεία. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει κάποιες εξηγήσεις στους εκλογείς μας. Γιατί καταργείται ένα δικαστήριο, γιατί καταργείται ένα ειδικό ειδικού τύπου δικαστήριο το οποίο ιδρύθηκε με βάση τις συνθήκες. Από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο δικαστήριο για κάποιους λόγους απέτυχε, θα έπρεπε να τους αναφέρουμε. Όχι τίποτα, Α, ξαφνικά αποφασίσαμε να το θάψουμε αυτό το δικαστήριο. Και αυξάνουμε έτσι απλά τον αριθμό των δικαστών ε, για το γενικό δικαστήριο. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν πολιτικές εξηγήσει και επειδή έχουν πολιτικές εξηγήσει έχουν και πολιτικές συνέπειες. Αυτό το οποίο θα πω λοιπόν τώρα εδώ είναι μια πολιτική παρατήρηση. Θα κάνω μια πολιτική παρατήρηση χωρίς καμία αμφιβολία για αυτό το οποίο θα πω. Έχουμε να κάνουμε με το μεγαλύτερο πολιτικό ψέμα στην λειτουργία της ευρωπαϊκής κοινότητας. Τι εννοώ εδώ. Ότι χρειάζονται περισσότεροι δικαστές για το Γενικό Δικαστήριο. Οι 28 δικαστές ήταν επαρκείς κάποτε. Γιατί θα πρέπει τώρα να διπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θέλουμε να τερματίσουμε τη λειτουργία του δικαστηρίου για τους υπαλλήλους και την εφαρμογή του υπαλληλικού κανονισμού. Ίσως υπάρχουν άλλοι, άλλες εξηγήσεις, εξηγήσεις για τις οποίες δυστυχώς συζήτηση δεν έγινε μέχρι τώρα καμία. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ με ε, ένα αριθμό σκοτεινών συμφερόντων δυστυχώς τα οποία δεν συζητάμε. Με τέτοιου τρόπου νοοτροπίες, με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο τρόπο άσκησης πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει πουθενά, δεν έχει μέλλον και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να υποκύψει στις επιθυμίες και τις, ε, ε, τις, ε, αυτά τα οποία θέλει να επιβάλλει το Συμβούλιο. Δεν έχουμε μέλλον δυστυχώς και είδαμε τι έγινε και στη Γερμανία. Ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντιευρωπαϊκό πνεύμα επεκτείνεται συνεχώς. Δεν έχει καμία εμπιστοσύνη ο εκλογέας απέναντι σε αυτούς οι οποίοι με συστηματικό τρόπο απονομιμοποιούν τα οικονομικά συμφέροντα, κυρίως τα οικονομικά επαναλαμβάνω συμφέροντα, των πολιτών. Δεν είναι θέμα αδικαϊκό, είναι θέμα εξουσίας, είναι θέμα πολιτικής και η πολιτική εξουσία στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνει προτάσεις και αποφασίζει εις βάρος του δικαίου, εις βάρος των εκλογέων, εις βάρος της δημοκρατίας. Λοιπόν, η πλειοψηφία το αποφάσισε, η ολομέλεια το αποφάσισε. Ας συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στο ψέμα Ας συνεχίσουμε εμείς ε, να κάνουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να πληρώνουν βαρύ τίμημα για τέτοιου είδους πολιτικές. Εγώ απέσυρα το όνομά μου από την έκθεση που είχα συντάξει γιατί η απόφαση την οποία πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα τεράστιο ψέμα και πάνω σε αυτό το ψέμα συνεχίζουμε να βασιζόμαστε δυστυχώς. Υπάρχουν άλλου είδους συμφέροντα τα οποία αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς, είναι συμφέροντα σκοτεινά, είναι συμφέροντα τα οποία ευνοούν αυτούς οι οποίοι δεν έχουν το θάρρος να υπερασπιστούν δημόσια τα συμφέροντά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δημιουργήσει ένα ειδικό δικαστήριο και το Κοινοβούλιο καταρχεί το δικαστήριο αυτό χωρίς να δώσει την παραμικρή εξήγηση. Δεν δόθηκε η παραμικρή εξήγηση για τον, για τον διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών. Έχουμε να κάνουμε τώρα δηλαδή με την πλήρη ανικανότητα α, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να ορίζει ένα αριθμό δικαστών διαφορετικό από τον αριθμό των χωρών μελών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε να κάνουμε τώρα όχι με ένα δικαστήριο αλλά με ένα σύνολο επιτρόπων που εξυπηρετούν εθνικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των αρμοδιοτήτων, του δικαίου, της δικαιοσύνης. Λοιπόν, δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Κυρία Ντελβό, έχετε το λόγο. Α, όχι, και ο κύριο Λεμπρετό. Σας, δεν σα έβλεπα γιατί έχει ήλιο. Ε, σας συγχωρώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο και να πω ότι δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον Μαρίνιο Πίντο σε αυτά τα οποία μόλις μας είπε. Είναι τεράστιο σκάνδαλο η κατάργηση του δικαστηρίου Νομίζω ότι σε νομικό επίπεδο η συνθήκη δεν το επιτρέπει πάρα πολύ απλά διότι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε δικαστικές δομές αλλά όχι να τις καταργήσουμε χωρίς τροποποίηση της συνθήκης. Σε πολιτικό επίπεδο είναι απαράδεκτο πολιτικά, άχρηστο πολιτικά να διπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών ε, εμείς κάναμε ακρόαση με τους Ευρωπαίους δικαστές και επιβεβαίωσαν την αντίληψη αυτή που είχαμε. Ο πραγματικός λοιπόν λόγος του διπλασιασμού αυτού θα πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι στις επίσημες εξηγήσει που δόθηκαν. Και αυτά ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πίντο. Ένα παιχνίδι σκοτεινών φαιών συμφερόντων. Σμικρίνεται ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ε, είμαι εδώ για να καταπολεμήσω αυτά που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα οποία βλέπω και ακούω ενισχύουν την αντίληψή μου εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε. Να κάνω και εγώ μία μία παρατήρηση. Θα ήθελα να πω ότι δεν είστε και τόσο ηλικιωμένος. Η κυρία Ντελβό. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι σέβομαι τις απόψεις όλων των βουλευτών. Ο καθένας από εμά είναι υπεύθυνο για αυτά τα οποία λέει, αλλά και ελεύθερος να τα πει. Εγώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι δεν είμαι υπέρ των συνωμοσιών. Θα ήθελα να πω ότι εγώ θέλω να εργαστώ υπέρ των συμφερόντων των ευρωπαϊκών εργάνων και να λειτουργήσουμε τη λειτουργία της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης συστατικό απαραίτητο για να αποκτήσει εμπιστοσύνη ο πολίτης στη λειτουργία της Ένωσης. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση που έγινε στο παρελθόν. Έχουμε μακρόν συζητήσει το θέμα της αναδιοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω να κλείσει η συζήτηση αυτή θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι για την αρμοδιότητα την οποία μπορεί να έχουμε για να καταργήσουμε το συγκεκριμένο αυτό ειδικό δικαστήριο. Ειδική φύσεως, επαναλαμβάνω, δικαστήριο. Το άρθρο 7 της συνθήκης, 57 ε, συγγνώμη, δίνει στους συνομοθέτες την δυνατότητα δημιουργίας ειδικής φύσεως δικαστικών οργάνων. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο οποίος έχει την αρμοδιότητα δημιουργίας έχει και την αρμοδιότητα κατάργησης. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ για το 257. Λοιπόν, αυτά πρόεδρε. Προτείνω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν να κλείσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Α, ο κύριος Πίντο ξαναζητάει το λόγο. Μικρόφωνο δυστυχώς δεν τον ακούμε εκτός μικροφώνου. Μία ερώτηση παρακαλώ θα ήθελα να θέσω. Ε, κυρία Ντελβό, μας είπατε ότι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί έχει και τη δυνατότητα να καταργεί νομικά. Έτσι είπατε. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω είναι πού βασίζεται αυτή την πρωτότυπη ερμηνεία. Αν γενικεύσουμε αυτή τη δικαϊκή αντίληψη θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι γονείς μπορούν να σκοτώσουν τα παιδιά τους. Αν γενικεύσουμε αυτή τη λογική όποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα όργανο μπορεί και να το διαγράψει, μπορεί και να το καταργήσει όποτε θέλει. Διέκοψα για να σας αφήσω να ακούσετε όλοι τους γέλοτες των συναδέλφων εδώ και να σεβαστώ το δικαίωμα να γελούν αυτοί που θέλουν να γελάσουν από αυτά τα οποία λέγω. Μπορείτε να γελάτε, ε, αυτό είναι έλλειψη σεβασμού απέναντι στους θεσμούς και γελιοποιείτε δημόσια αυτό το οποίο είπα. Προσπαθώ να είμαι σοβαρός και προσπαθώ να τονίσω αυτά τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σοβαρά. Και γι' αυτό λοιπόν τέτοιου είδους δυνατοί γέλοτες είναι σαφέστατα δείγμα έλλειψης σεβασμού. Απαξιώνεται με πρωτόγονο τρόπο αυτό το οποίο είναι ε, ε, δικαίωμα κάθε συναδέλφου να λέει. Έχετε καθήκον και υποχρέωση να ακούτε με σεβασμό αυτά τα οποία λέγουν οι συνάδελφοι μάθετε να ακούτε. Είναι η πρώτη λειτουργία του βουλευτή. Λοιπόν κυρία Ντελβό, ξανά η ερώτησή μου. Πού βασίζεται την ιδέα αυτή ότι όποιος δημιουργεί μπορεί και να καταστρέφει. Είπατε ότι αυτός ο οποίος δημιουργεί ένα όργανο έχει το δικαίωμα να το καταργήσει. Σε ποιο επίπεδο νομικής τεκμηρίωσης ανάγεται τη συγκεκριμένη ερμηνεία. Σας εξήγησα, σε αυτή την περίπτωση αν αποδεχθούμε μια τέτοιου είδους αντίληψη τότε δεν είμαστε μακράν της αναγνώρισης του δικαιώματος θανάτωσης αν είμαστε υπεύθυνοι για την δημιουργία και τη γέννηση ενός προσώπου. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η αντίληψη η οποία τεκμηριώνει την κατάργηση του δικαστηρίου είναι απαράδεκτη και μιλάμε για ένα πρόσφατο δικαστήριο κυρία Ντελβό. Γιατί καταργείται κυρία Αντελβό, δεν υπάρχουν εξηγήσει. Έγινε κανένα σοβαρό λάθος σε σχέση με το όργανο αυτό. Είναι ένα όργανο το οποίο δημιουργήθηκε από τις συνθήκες. Γιατί κάτι το οποίο προβλέπεται από τις συνθήκες θα καταργηθεί εκτός συνθήκων από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε αυτό. Οι προτάσεις τις οποίες κάνετε λυπάμαι αλλά δεν είναι τεκμηριωμένες και οι πολίτες δεν θα τις κατανοήσουν. Βοηθήστε τους πολίτες λοιπόν να κατανοήσουν, βοηθήστε με εμένα να κατανοήσω. Και επαναλαμβάνω, εγώ ακούω όλο τον κόσμο με τον μέγιστο ε, θεμασμό και αυτά τα οποία άκουσα από πλευράς της κυρίας Χάουταλα και τα λοιπά νομίζω ότι είναι ανάξια του πολιτικού της κόμματος και ανάξια της ε, σοφής και ε, επιβαλόμενης συμπεριφοράς ενός κοινοβουλευτικού. Κοιτάξτε κυρία Χάουταλα θα πάρει το λόγο. Θα ήθελα όμως να σας πω εδώ ότι όλοι ε, όλοι εξεπλάγησαν από το εύρος της αναλογίας την οποία χρησιμοποίησατε και ιδιαίτερα τώρα πρωί πρωί να ακούμε τέτοια πράγματα ε, μας ε, εξέπληξαν. Αλλά τα επιχειρήματά σας είναι σεβαστά. Κύριε Πρόεδρε, είπατε αυτά τα οποία θα ήθελα να πω. Το θέμα δεν ε, ήταν αυτό το οποίο με έκανε να αντιδράσω έτσι, δεν είναι η ερμηνεία του 257. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και δεν θέλω εγώ να φανεί ότι γέλασα για κάποιον μόνο και μόνο έχει διαφορετική άποψη. Απλά η αναλογία την οποία ανέφερε ο, ο κύριος Πίντο με εξέπληξε. Η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση, λέει η κυρία Ντελβό δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε μία ενιαία άποψη σε σχέση με το αν το 257 επιτρέπει ή όχι την κατάργηση του δικαστηρίου. Νομίζω ότι οι νομομαθείς ανάμεσά μας, οι εξειδικευμένοι νομομαθείς, θα μπορούσαν να εκφέρουν την άποψή τους. Εγώ πάντως προτείνω να κλείνει η συζήτηση, να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Το έχουμε συζητήσει ώρες ολόκληρες ε, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό αναλυτικά, όχι γιατί θέλουμε να τιμωρήσουμε το συγκεκριμένο δικαστήριο, αλλά γιατί πάρα πολύ απλά θεωρήσαμε ότι προς όφελος της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γενικότερα και των επιμέρους συνιστοσών του από την άλλη, θα έπρεπε να υπάρξει μια συγχώνευση των δικαστικών κοινοτικών οργάνων. Λοιπόν, η απόφαση έχει ληφθεί, θυμίζει ο Πρόεδρος. Εμείς μιλάμε για την εφαρμογή της απόφασης. Σας ευχαριστώ όλους. Βλέπω ότι ήδη από, από πρωίας υπάρχουν έντονες αντιλήψεις για τα πράγματα. Το επόμενο θέμα είναι θέμα της κυρίας Χάουταλα. Έχετε το λόγο κυρία Χάουταλα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η αιτήσια, το ετήσιο σχέδιο έκθεσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Βασίζεται στην έκθεση της Επιτροπής του 2014 και βλέπω εδώ με χαρά τον εισηγητή από πέρσι, τον κύριο Χρυσόγονο. Η εφαρμογή του δικαίου, η συμμόρφωση είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Περιμένουμε γνωμοδοτήσεις και άλλων επιτροπών, αλλά εμείς θα καταρτήσουμε την έκθεση και θα την υποβάλουμε στην Ολομέλεια. Ως φετινή εισηγήτρια έχω ετοιμάσει ένα σχέδιο και περιμένω τις απόψεις σας, νέες ιδέες, ενδεχομένως που εγώ δεν έλαβα ακόμη υπόψη. Αναφέρω θέματα γύρω από τρεις τομείς κυρίως. Καταρχήν το EU Pilot. Δεύτερον, η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και σε χώρες ένταξης ή ε, σύνδεσης, που είναι δύσκολο θέμα, και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου που θα πρέπει να ενδυναμωθεί μέσα από αποτελεσματικότερη διοίκηση. Τώρα, για το ε, EU Pilot και τους σχετικούς φακέλους, η έκθεση δείχνει ότι το περιβάλλον, οι μεταφορές, η εσωτερική αγορά είναι οι τομεί όπου γίνονται οι περισσότερε παραβιάσει που έγιναν το 2014. Η ετήσια έκθεση τη Επιτροπή τονίζει επίση ότι ο αριθμό των επίσημων διαδικασιών επί παραβάση ε, μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι βασικό. Σύμφωνα με την Κομισιόν, αυτό δείχνει την αποτελεσματικότητα του διαλόγου με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της διαδικασίας EU Pilot. Τώρα, νομίζω ότι έχουμε λόγο να παραμένουμε επιφυλακτικοί, γιατί το Κοινοβούλιο δεν έχει πρόσβαση σε όλα αυτά, στον, στον διάλογο αυτό και σε εκκρεμείς υποθέσεις. Ένα συμπέρασμα που μπορεί να συναχθεί λοιπόν είναι ότι η επιβολή του ενωσιακού δικαίου ακόμη δεν είναι αρκετά διαφανής. Και σίγουρα ένας τρόπος βελτίωσης της εφαρμογής του νόμου είναι η ανάπτυξη της διοίκησης της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο αυτό πολλές φορές έχει ζητήσει συνεκτικότερη προσέγγιση και ε, σε λίγο θα το επαναλάβει αυτό όταν υποβάλει το κείμενο κανονισμού στην Κομισιόν για ανοιχτή και ανεξάρτητη και δημόσια ε, ε, διοίκηση της Ένωσης. Η ομάδα εργασίας τώρα έχει παρουσιάσει ένα πιο ουσιαστικό όνομα για το κανονισμό. Θα υπάρχουν πρότυπα για την κοινοποίηση, ε, χρονικά περιθώρια, υποχρέωση αιτιολογημένης γνώμης και ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση στο φακελό του. Ε, αν θέλουμε να δυναμώσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, πρέπει να ε, δυναμώσουμε και τη σωστή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Έτσι ήθελα να ε, εστιάσουμε τις προσπάθειες ούτως ώστε να έχουμε μια ανεξάρτητη αποτελεσματική ανοιχτή διοίκηση. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στα υφιστάμενα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς οι χώρες ένταξης, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες βέβαια είναι στα Δυτικά Βαλκάνια, και οι χώρες με τις οποίες υπάρχουν συμφωνίες σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αυτές συμμορφούνται με το νοσιακό δίκαιο. Θυμίζω ότι τρεις χώρες σύνδεση είναι η Ουκρανία, η Γεωργία και η Μολδαβία. Έφυστο την προσοχή στην ανάγκη να τους στηρίξουμε καταλήλως για να συμμορφούνται με το νοσιακό δίκαιο και να το εφαρμόζουν σωστά. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει πολύ σοβαρό έργο εδώ, ενθαρρύνοντας και ενδυναμώνοντας την κατανόηση ε, από τα κοινοβούλια αυτά του πώς μεταφέρονται ε, που ενταφέρεται το ενωσιακό δίκαιο μετά το Πάσχα, μια μικρή αντιπροσωπεία που είναι ακόμα ανοιχτή για να έρθουν και άλλα μέλη, θα πάνε για τριήμερο στη Γεωργία για να δουν πώς εξελίσσεται το έργο αυτό σε αυτή τη χώρα και εδώ συνεχίζεται λίγο η καλή εμπειρία μας μιας ε, αποστολής στην Ουκρανία μαζί με την Ίντα. Και ήταν η προσωπία ίντα εκεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία για να εφαρμόσει τη Συμφωνία Σύνδεσης. Αυτά έχω καταγράψει. Ξέρω ότι άλλοι συγητές άλλων ετών έδωσαν έμφαση σε άλλα θέματα. Είμαι όμως ανοιχτή στις ιδέες και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία εισηγήτρια. Η κυρία Κόφμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια που θεωρώ ότι ετοίμασε ένα καλό σχέδιο έκθεσης το οποίο μπορώ και να στηρίξω. Μόλις τώρα τόνισε ότι της είναι σημαντικό ότι το Κοινοβούλιο δηλαδή κατά την ανάλυση της στήρησης του ενωσιακού δικαίου θα πρέπει να περιλάβει και άλλες χώρες με συμφωνίες σύνδεσης και τις χώρες ένταξης. Εγώ το προσυπογράφω αυτό με μεγάλη θέρμη. Πιστεύω ότι είναι σωστό και απαραίτητο σε αυτή τη διαδικασία ως Κοινοβούλιο να συμμετέχουμε και εμείς. Επίσης θετικό είναι ότι η εισηγήτρια εντοπίζει το θέμα της στενότερης συνεργασίας Κοινοβουλίου Κομισιών και την καλύτερη πρόσβαση του Κοινοβουλίου στη διαδικασία EU Pilot και τις διαδικασίες επί παραβάση. Είναι σημαντικά αυτά και στηρίζω επίσης και το αίτημά της για μια νομοθετική πρόταση της Κομισιόν για μια διαδικασία ευρωπαϊκού ε, διοικητικού δικαίου. Θα ήθελα να αναφέρω και ορισμένα άλλα θέματα. Πιστεύω ότι αυτή η ετήσια έκθεση είναι και κομμάτι του τωρινού θεματολογίου της Κομισιόν για την καλύτερη νομοθεσία. Θα θυμάστε ότι την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, είδαμε και εγκρίναμε τη νέα διοργανική συμφωνία και ίσως σε σχέση με αυτή την συμφωνία θα πρέπει να δούμε μήπως ε, μπορεί στην έκθεση να συμπεριληφθούν κάποια καινούργια στοιχεία. Παράδειγμα, ε, υπάρχει μια τροπολογία ε, που ήθελα να υποβάλω ότι θα πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη-μέλη ε, αν θέλουν ρύθμιση πέραν μιας οδηγίας. Ε, αν αποφασίσουν δηλαδή να προσθέσουν κάτι ακόμα. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντική καινοτομία γιατί καμιά φορά οι πολίτες δεν ξέρουν αν πρόκειται για ευρωπαϊκή νομοθεσία ή τι έχει προσθεθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία στο εθνικό πια επίπεδο. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν ποιος φέρει ευθύνη για ποιο πράγμα και αυτή την καινοτομία πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας στην εφαρμογή του ε, νοσιακού δικαίου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγωνος. Thank you, Chairman. I admire very uh, Ευχαριστώ. Πολύ θαυμάζω τη διπλωματική διατύπωση της εισηγήτριας, ότι δηλαδή το Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει πιο διαρθρωμένο ρόλο και να εξετάζει την συμμόρφωση των υποψηφίων χωρών προς το ενωσιακό δίκαιο. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν υποψήφιες χώρες που δεν συμμορφούνται με το ενωσιακό δίκαιο και όχι μόνο δεν συμμορφούνται με βασικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, ιδιαίτερα ε, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου και της δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν υποψήφιες χώρες ε, που αντί να επιτελούν πρόοδο σε αυτούς τους τομείς, αντίθετα υπο... επιδεινώνονται κάθε χρόνο. Και το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο παράδειγμα είναι η Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο την ανέχεται, αλλά και την ενθαρρύνει. Ενθαρρύνει το καθεστώς Ερντογάν στην παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ιδιαίτερα της κουρδικής μειονότητας, αλλά και του τουρκικού λαού συνολικά. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην ελευθεροτυπία, την ελευθερία λόγου κλπ. Τους ενθαρρύνομαι λοιπόν να συνεχίζουν προς αυτή την κατεύθυνση λόγω πολιτικών στόχων και σκοπιμοτήτων. Φαίνεται ότι είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε από τις αρχές μας όλο και περισσότερο γίνεται αυτό. Ε, συν το χρόνο. Και αυτό αποτελεί λόγο ανησυχίας για μένα. Και όχι μόνο για μένα υποθέτω, αλλά για πολλούς ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίφσκα. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χαουτάλα για αυτό το σχέδιο κειμένου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να τονίζουμε τη σημασία διαφόρων ζητημάτων ε, στις εκθέσεις μας και αυτό λειτουργεί αρκετά καλά. Η δουλειά σας είναι πολύ καλή. Θέλω να ευχαριστήσω τους προλαλήσαντες γιατί αναφερθήκαν σε πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία και εγώ θα ήθελα να τονίσω. Μιλούμε με όμορφα λόγια, στη συνέχεια όμως η εφαρμογή είναι κάπως προβληματική. Πολύ συχνά οι πολίτες εξαπατώνται από τις δικές τους εθνικές αρχές, κρατικές αρχές, οι οποίες λένε στον κόσμο «Μα αυτά περιμένουν από μας οι Βρυξέλλες». Σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και πολύ συχνά τα προβλήματα προκύπτουν από το εθνικό επίπεδο ενώ το ανάθεμα ρίχνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να παρεπονεθούμε γι' αυτό. Και θα έπρεπε να αναδείξουμε την ευθύνη που φέρει το εκάστοτε επίπεδο διοίκησης, εντός και εκτός. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε εκθέσεις για το πόσο έχει προοδεύσει κάθε χώρα στην ενσωμάτωση του κοινοτικού και εκτιμένου. Ε, συμφωνώ με αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει πρόοδος στις υποψήφιες χώρες. Είναι τεράστια η προσπάθεια που απαιτείται. Πριν από το 2004 στην Πολωνία, ο κόπος που καταβάλαμε ήταν τεράστιος. Ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά από πλευράς κυβέρνηση να ενσωματώσει όλο το ενωσιακό κεκτημένο όταν η Πολωνία ήταν υποψήφια χώρα. Θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν για την πρόοδο τη κάθε χώρα να υποβάλλονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. πρόοδος ε, στο ενωσιακό δίκαιο που έχουν σημειώσει υποψήφιες χώρες ή ε, οι συνδεδεμένες χώρες. Και τέλος, ως προς τη διοργανική συμφωνία, την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είπα ότι είναι μια συμφωνία η οποία υιοθετείται μόνο μία φορά στο τόσο. Πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να υιοθετηθεί ξανά τέτοιου είδους συμφωνία. Απ' την άλλη πλευρά, η ποιότητα του ενωσιακού δικαίου θα πρέπει να είναι κύριο μέλημά μας καθημερινά. Επομένως, η Συμβουλή προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τουλάχιστον προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να εκτιμήσουν ιδιαίτερο τη δουλειά της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Είμαστε μια πολύ σημαντική επιτροπή, ενδεχομένως η σημαντικότερη από τις μικρές. Και θα πρέπει το έργο μας, η δουλειά μας, να παρουσιάζεται στην Ολομέλεια σε ένα εύλογο χρονικό ε, διάστημα και την κατάλληλη χρονική στιγμή, όχι 11 και το βράδυ τη νύχτα αλλά σε συνεδριάσεις όπου συζητώνται ε, πολύ σημαντικά νομικά θέματα μεγάλου βεληνικούς. Αυτό θα πρέπει να ζητούμε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Κυρία Χαουτάλα, αν δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, σας παρακαλώ να τον πάρετε εσείς. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι η έκθεση θα γίνει συλλογικό έργο της Επιτροπής και ευχαριστώ όλες τις απόψεις από τους συναδέλφους Κάουφμαν, Χρυσόγονο, Σίφκα. Νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνουμε λίγο σε αυτή την ιδέα ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει και να ενημερώνεται περισσότερο ε, πάνω στα στάδια μεταφοράς και εφαρμογής του ενωσιακού κεκτημένου στις χώρες σύνδεσης και ένταξης. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι που ο κύριος Χρυσόγονος έθεσε ένα πάρα πολύ θεμελιώδες ζήτημα και ε, ε, ίσως ήμουν υπερβολικά διπλωματική πραγματικά, αλλά είναι αλήθεια, δεν μπορεί να μεταφέρει στο νοσιακό και εκτιμένο στον τομέα της πολιτικής μεταφορών ή προστασίας των καταναλωτών αν δεν έχεις ε, στέρεα θεσμούς, αν δεν ισχύει το κράτος δικαίου, αν δεν έχεις διάκριση εξουσιών, αν έχεις διαφθορά και αν δεν έχεις διαφάνεια. Λοιπόν, είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, όχι μόνο στην Τουρκία που είναι ίσως το πιο εξέχον παράδειγμα αλλά υπάρχουν παρόμοια θέματα και σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες ένταξης και σύνδεσης και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Ευχαριστώ για τη διπλωματική παρατήρησή σας, για την δική μου υπερβολικά διπλωματική διατύπωση. Και ε, όντως ε, πρέπει να προσθεθούν κάποιες παράγραφοι για την εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για την Καλύτερη Νομοθεσία, αν και γνωρίζω ότι θα υπάρξει έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας μαζί με την ΑΦΚΟ και την Επιτροπή μας. Αλλά παρόλα αυτά ναι, να το εντάξουμε και εδώ και η κυρία Κάουφμαν και ο κύριος Ζήφκα ανέφεραν το θέμα του gold plating, αυτού του κανονιστικού υπερθεματισμού, ε, που παραπλανά τους πολίτες. Και τέλος, είναι καλό κάθε χρόνο να θέτω με κάποιο θέμα. Πέρσι ο κύριος Χρυσόγονος εστιάστηκε επιτυχώς στο θέμα των πολιτικών λιτότητας. Ε, ως παραβιάσεις, δηλαδή η υπερβολική ε, λιτότητα παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και νομίζω ότι η χώρα του πέρασε πολλά ε, εδώ. Πριν καταθέσουμε τις τροπολογίες θα συνεννοηθούμε βέβαια και από πριν θα είμαστε σε επαφή για να προλάβουμε και τις γνώμες των άλλων επιτροπών, της νομοδοτήσεις. Ε, υπάρχει ήδη κάτι από την Επιτροπή Απασχόλησης, αν δεν κάνω λάθος, και είναι περίεργη κάπως πρόταση μια, ότι μια σημαντική επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει υποεπιτροπή για να, είναι, για να παρακολουθεί την εφαρμογή του νοσιακού δικαίου. Δεν μου φαίνεται ότι είναι και τόσο καλή πρόταση, αλλά θα τη δούμε συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, το 9 αναβάλλεται. Και εσείς έχετε το λόγο πάλι, κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες είναι, θα έλεγα, μία από τις πιο πρόσφατες και τις πιο σύγχρονες συμβάσεις που πράγματι μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες σε όλο τον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως η οποία έχει κυρώσει αυτή τη σύμβαση Και υπάρχει αυτή η Επιτροπή η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή ε, τη σύμβαση του ΟΗΕ, στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Η γνωμοδότηση αυτή υποβάλλεται λοιπόν στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και οφείλω να πω ότι ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων επιτροπών εισηγητών είναι πολύ καλός. και η σχετική ομάδα εξέταση θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρίες είναι, εμπλέκεται σε αυτές τις συζητήσεις και είναι πολύ δραστήρια. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι Αυτό που χρειάζεται είναι να τονίσουμε τα εξή, ότι η Επιτροπή θα αναθεωρήσει το σύνολο ε, της ε, κοινοτικής νομοθεσίας για να διασφαλίσει ότι συνάδει με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Οφείλουμε να έχουμε μηχανισμούς ε, προσφυγής που, για τα άτομα με αναπηρίες σε σχέση με την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους έτσι όπως προβλέπονται στη σύμβαση του ΟΗΕ και να μεριμνήσουμε να αρθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες εξαιρέσεις για ε, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, copyright κτλ. Ε, πράγματα τα οποία δεν είναι αντίθετα με τη συνθήκη του Μαρακές που επίσης μας ε, απασχολεί και είμαστε αρμόδιοι ως Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ο Μαξ Άντερσον είναι ο εισηγητής για το σχετικό θέμα. Εκφράζω τη λύπη μου διότι το Συμβούλιο συζήτησε την απλούστευση της πρόσβασης δημοσίων εγγράφων για τους πολίτες στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αθέμα αρμοδιότητας της Μαντιντελβό, δεν επέκτηνε το πεδίο εφαρμογής ε, στην πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες. Και εκφράζω τη λύπη μου γι' αυτό. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή θα είναι σύντομη θα είναι τα θέματα πολύ πιο ε, ε, περιεκτικά στην Επιτροπή Απασχόλησης και Νομικών Υποθέσεων. Εμείς δεν έχουμε και πολλά να πούμε, ε, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια και παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιος άλλο το λόγο, να δώσω το λόγο στην κυρία Ντελβό. Και εγώ θα ήθελα να εξηγήσω το εξής. Όταν ζητήσαμε τα πιστοποιητικά για αναπηρίες, οι βεβαιώσεις δηλαδή αναπηρίας ε, να μπουν ε, στα έγγραφα που γίνονται αποδεκτά ως δημόσια έγγραφα δεν υπήρχαν αντιρρήσεις, αλλά αφού δεν υπήρχαν στην αρχική πρόταση, η Επιτροπή είπε ότι πρέπει να κάνει αξιολόγηση και παρακολούθηση για το ποιες θα ήταν οι συνέπειες του να συμπεριληφθούν αυτά. Επομένως στην έκθεση υποσχέθηκε η Επιτροπή ότι θα κάνει την αξιολόγηση για το ποιες συνέπειες θα έχει εάν οι βεβαιώσεις αναπηρίες θεωρούσαν, θεωρούνται ως έγγραφα που εντάσσονται στα δημόσια κτλ. Δύο χρόνια πέρασαν. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν κατά. Ε, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Για λόγους τυπικούς δεν ήταν σε θέση να δεχτούν, να συμπεριληφθεί κάτι που δεν είναι στην αρχική πρόταση, χωρίς να έχει γίνει πρώτα ε, μελέτη αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών. Και γι' αυτό δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής. Ευχαριστούμε την κυρία Ντελβό, ο κύριος Μαρίνιο Πίντο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στις αναπηρίες, στα άτομα με αναπηρίες και στα δικαιώματά τους και κυρίως να σχολιάσω δύο ή τρία σημεία. Καταρχάς να πω ότι τίνουμε να έχουμε ανθρωπιστικό δίκαιο συμβολικό. Στα νομικά κείμενα απαριθμούμε όλα τα δικαιώματα, όμως στη συνέχεια στην πρακτική άσκηση των δικαιωμάτων κάνουμε πολύ λιγότερο για να μην πω ότι δεν κάνουμε και τίποτα απολύτως. τα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, τα ανθρωπιστικά δικαιώματα είναι αυτά για τα οποία γίνονται ε, μεγάλες ρητορίες, δηλώσεις πομπόδης και ε, έχουμε πάρα πολύ καλή διατύπωση και πλούσια στο αιτιολογικό, ε, στα εκτιμόντες στις αιτιολογικές σκέψεις. Στη συνέχεια όμως δεν γίνεται και πολλής λόγος. Θα ήθελα να μιλήσω για τα άτομα που έχουν διανοητική αναπηρία και για το πρόβλημα της ψυχικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ήμουν φοιτητή, έλεγαν ότι ο τρελός είναι αυτός που έχει χάσει τα πάντα εκτός από, το δίκιο του και από τη λογική του. Ε, και θέλω να σας ευχηστήσω την προσοχή ακριβώς σε αυτό το θέμα. Στην Πορτογαλία κάποιος που πάσχει από διανοητική αναπηρία δύναται τελικά να κρατηθεί, να είναι υποκράτηση σε όλη του τη ζωή χωρίς να έχει θεωρηθεί ένοχος ή χωρίς να έχει διαπράξει οτιδήποτε. Μόνο και μόνο επειδή αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί κάποιο κίνδυνο. Ο Πορτογαλικός νόμος για τη διανοητική, για τη ψυχική υγεία προβλέπει ε, ε, εξοφίτσιο εγκλισμό του, του ε, προσώπου χωρίς να έχει διαπράξει ποτέ καμία, κανένα αδίκημα ποινικό. Ένας όμως ε, εγκληματίας θα πρέπει να έχει διαπράξει κάτι που να ορίζεται ξεκάθαρα από τον κώδικα ποινική δικονομίας για να διαταχθεί η κράτησή του η στέρηση της ελευθερίας του, ο περιορισμός του. Ένας όμως που πάσχει από ψυχική υγεία κρατείται χωρίς να έχει διαπράξει τίποτα σε ε, εδρήματα τα οποία είναι βέβαια νοσοκομεία αλλά ουσιαστικά είναι και φυλακές. Θεωρώ ότι πρόκειται για καταστρατήγηση ανθρώπινων δικαιωμάτων και μάλιστα ενός ατόμου το οποίο δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το οποίο δεν δύναται να τα ασκήσει ε, εν ορθό το λόγο διότι δεν έχει την ικανότητα να το κάνει και καταστρατηγούνται και καταπιατούνται τα δικαιώματά του. Και για να συνδέσω αυτά θέλω να εκφράσω από τη συμφωνία μου με τον κύριο Χρυσόγονο όσον αφορά στη νομοθεσία ορισμένων χωρών οι οποίες αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις μετοχές τους να έχουν ανέβει πάρα πολύ ε, για λόγους πολιτικού οπορτουνισμού. Σύμφωνα απολύτως λοιπόν με αυτά και θέλω οι, οι, οι πάσχοντες να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους α, οι υπολείπους και να ενισχύσουμε ακριβώς την προστασία τους, γιατί οι ίδιοι δεν δίνανται να τα ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Κομοντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδη εισηγήτρια για την ίδια έκθεση στην Επιτροπή Κουλ του Πολιτισμού και συμφωνώ μαζί σας κυρία Χαουτάλα. Είναι πολύ καλή η συνεργασία μεταξύ των εισηγητών, των σκιωδών εισηγητών και ούτω καθεξής με τους αντίστοιχους ε, συναδέλφους αρμοδίους στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αν διαβάσει κανείς το πόρισμα της Επιτροπής του ΟΙΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σύμβαση αυτή, και αν αυτό το συνδέσει με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων τη δική μας, νομίζω ότι τρεις είναι οι τομείς που μας αφορούν και τους καλύψατε. Ότι δηλαδή η Επιτροπή παραπονεί παραπονιέται γιατί δεν κάνουμε mainstreaming ε, στα ατομικά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, το οποίο λέτε και σωστά. Περιμένει η Επιτροπή του ΟΗΕ να το πράξουμε. Ότι δηλαδή η διάσταση της αναπηρίας να αναλυθεί σε κάθε ευρωπαϊκό νομοθέτημα και το τρίτο που έχω εντοπίσει είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει ένα σύστημα διασφάλιση έτσι ώστε να δει ότι πράγματι αποτελεσματικά εφαρμόζεται η σύμβαση από τα κράτη-μέλη. Πράγματι μπορεί να έχει ενσωματωθεί στο κοινοτικό κεκτημένο ή στο εθνικό ε, ε, ε, κεκτημένο Μία από τις συστάσεις όμως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεριμνήσει για να επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν επαρκείς δομές στα κράτη-μέλη για να εφαρμοστεί σωστά η σύμβαση του ΟΗΕ. Θα έλεγα λοιπόν ότι εμέσως εμείς ως Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πέρα από όλα αυτά μπορούμε να ζητήσουμε και το εξής. Κάθε φορά που δίδεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να βεβαιωνόμαστε ότι έχει γίνει mainstreaming της διάστασης της αναπηρίας γιατί έχει υπάρξει χρηματοδότηση ευρωπαϊκή και για project συγκεκριμένα, έργα συγκεκριμένα για αναπηρία, η οποία χρηματοδότηση όμως τελικά δεν επέφερε τις αλλαγές που θέλαμε. Αντί να υπάρχει ένταξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο, ουσιαστικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έγινε περισσότερη γετοποίηση των ατόμων με αναπηρίες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ας πούμε το χτίσιμο ενός σπιτιού για άτομα με αναπηρίες οι οποίοι θα ζούσαν εκεί πέρα και τελικά άτομα με αναπηρίες στηβάζονται σε αυτές τις κατοικίες και σε αυτά τα κτίρια που είναι μόνο για άτομα με αναπηρίες, δηλαδή δημιουργούνται μικρά γκέτο. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία μας δεν συνεχίζει να κάνει διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες. Να διασφαλίσουμε επίσης ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να στηρίζουν σχέδια και έργα που συνάδουν με την πολιτιστική αλλαγή, την αλλαγή νοτροπίας ε, την οποία, στην οποία αποσκοπεί η σύμβαση του ΟΗΕ. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ. Θέλετε να παρέμβετε. Παρακαλώ, εσείς, κυρία μου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους παρόντες. Πράγματι είναι πολύ σημαντική αυτή η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και για μας και για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αναφερθήκατε στη συνθήκη του Μαρακές, ε, κάτι το εξίσου σημαντικό. Να σχολιάσω κάποιες παρατηρήσεις που έγινα. Η Επιτροπή εργάζεται, είναι πολύ ενεργή, ε, όχι μόνο στις αναπηρίες, τα άτομα με αναπηρίες για την αποϊδρυματοποίησή τους και χρηματοδοτή τι διάφορα έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, έργα με στόχο την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρίες και στο προγραμματικό πλαίσιο 2014-2020 υπάρχουν οι προϋποθέσεις εξάντε, εκ των προτέρων δηλαδή, για τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα στα κράτη-μέλη, ε, όταν δηλαδή λαμβάνονται υπόψη τα άτομα με αναπηρίες. Ε, έργα για την αποϊδρυματοποίηση στα κράτη-μέλη. Είναι ένα έργο περίπλοκο, μακρόχρονο, δύσκολο. Εξετάζουμε λοιπόν αυτά τα project και έτσι τα περνάμε από κόσκινο και στην ενδιάμεση αναθεώρηση της προγραμματικής περίοδου μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό ε, για το πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη. Σημείωσα επίσης ότι Πράγματι, οι ψυχικώς πάσχοντες είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματοδοτούμε μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την ε, διανοητική αναπηρία, με τους ψυχικώς πάσχοντες. Πάρα πολλά μένουν να γίνουν, συμφωνώ και γι' αυτό κάθε είδους συμβολή και συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μας βοηθήσει. Θα δουλέψουμε ακόμα καλύτερα και ακόμα περισσότερο και με την Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών και με τα κράτη-μέλη. Ναι, εγώ έχω ερώτηση, μια ερώτηση. Ποιος ελέγχει την σωστή χρήση των κονδυλίων που διανέμεται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ρωτάει ο Πρόεδρός σας. Απάντηση. Δίνουμε grants, επιδοτήσεις, ενισχύσεις για τη λειτουργία τους. Αυτό γίνεται με διαγωνισμό, με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Έτσι χρηματοδοτούμε και ε, ε, έχουμε ελεγκτές και ε, γίνεται δημοσιονομικός έλεγχος και συντάσσονται εκθέσεις για τα κονδύλια που ε, δίνουμε 9 εκατομμύρια σε 8 μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Χρηματοδοτούμε τα σχέδια της δραστηριότητας. Επομένως, λέει ο πρόεδρος, ε, τα χρήματα δίδονται αναέργο. Υπάρχει project, ναι. Ε, υπάρχει ένας διαγωνισμός τριετούς έκτασης χρονικής. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις υποβάλλουν ένα σχέδιο δράσης, ένα πρόγραμμα εργασιών με δραστηριότητες πολύ συγκεκριμένες και κάνουμε την αξιολόγηση κάθε δραστηριότητα σε αιτήσια βάση μια πολύ εκ παρακολούθηση της εφαρμογής. Βεβαίως είναι αυτό δικητικά επαχθές και ε, γραφειοκρατικό. Μπορεί να έρθει η δική εμπειρογνώμων εδώ να σας ενημερώσει περισσότερο. Δεν είναι εύκολο να αποδώσουμε πάντοτε λογαριασμό. Ούτε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι εύκολο να αποδίδουν λογαριασμό γιατί δεν έχουν ούτε αυτέ τη γιγάντια διοικητική δομή που χρειάζεται. Και προσπαθούμε να του διευκολύνουμε. Βέβαια, αυτό όμω είναι ο ένα έλεγχο και ο άλλο έλεγχο είναι ο τεράστιο έλεγχο που γίνεται στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η Επιτροπή ε, ε, κάνει απολογισμό των κονδυλίων που έχουν χρησιμοποιηθεί κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Η Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση συντάσσει ετήσια έκθεση πολύ ουσιαστική και εκεί απαριθμεί λεπτομερώ τι έχουν γίνει τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το ελεκτικό συνέδριο μα ελέγχει, αλλά και έχουμε και ad hoc ελέγχου ε, έκτακτους και έχουμε και εσωτερικό μηχανισμό στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη αξιολογούν επίσης τα έργα και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυτό το μηχανισμό επιτήρηση. Όλα αυτά είναι καινούρια, ε, αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή, εξελίσσονται και έτσι έχουμε και εμεί το feedback, την τροφοδότηση από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει επί τη βάση των εμπειριών του. Ευχαριστούμε, λέει Κυρία Χαουτάλα, τα συμπεράσματά σα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Μάριο Πίνιο και την αμέλεια που δείξαμε προς ε, την ψυχική νόσο. Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δέκα χρόνια έκανε βελτιώσεις, γιατί όταν μιλάμε για δημόσια υγεία και η ψυχική υγεία είναι σημαντικό κομμάτι αυτής γιατί είναι πηγή πολλών προβλημάτων και αποκλεισμού από την κοινωνία. Αλλά ε, συνάγω από αυτό που είπε ο κ. Μαρίνιο Πίντο ότι υπάρχει πολύ έμεση διάκριση, υπάρχουν έμεσες διακρίσεις, αν όχι και άμεσες διακρίσεις στην αντιμετώπιση των ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα. Ίσως αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε πιο λεπτομερώς. Όλοι οι άλλοι ομιλητές ε, είπαν σωστά πράγματα. Κυρία, κυρία Κομοντίνη, ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε και για την πολιτισμική αλλαγή που θα επιφέρει, όπως υποθέτουμε αυτή η σύμβαση και πρέπει να δούμε ε, τι δομές ε, υπάρχουν για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων νομοθετικών αλλαγών και στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν είναι η Επιτροπή μας που πρέπει να δει το πώς θα ε, χρησιμοποιηθούν ενωσιακά κονδύλια για την ε, ενσωμάτωση της αναπηρίας σε όλες τις χρηματοδοτήσεις. Πάντως σίγουρα το Κοινοβούλιο πρέπει να το κοιτάξει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μου επιβεβαιώνει ότι τα συμπεράσματα της Επιτροπής ε, για τη Σύμβαση είναι σημαντικά για την Κομισιόν και βέβαια ε, υπάρχει ε, και ένα θετικό όφελος από την ενθάρρυνση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο σημείο 12. Το σημείο 11 το οποίο μας αφορά και αφορά και την κυρία Περζερό και την κυρία Ρεντά, αλλά και εσάς κυρία Χαουτάλα. Ένα σύντομος απολογισμός της ε, αποστολής στην Ουτρέχτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου. Ξεκινάτε εσείς κυρία Μπερζερό. Μου άρεσε πολύ αυτό το ταξίδι, αυτή η αποστολή στην Ουτρέχτη. Ευχαριστώ τους ε, διοργανωτές και με ενδιαφέρει ιδιαίτερος για λόγους ε, πολύ βασικούς και αρχικούς να επισκεφθώ το Διαιτητικό Δικαστήριο το, για το οποίο είχα ακούσει τόσα πολλά όταν έκανα το διδακτορικό μου για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό ήταν ε, ένα όνειρο για μένα και συνειδητοποίησα ότι αυτός ο οργανισμός ο οποίος δουλεύει με ε, πολύ ε, αξιόλογους νομικούς, είναι ε, πολύ ενδιαφέρον οργανισμός και μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για το διεθνές δίκαιο. Και παρόλο που υπάρχει διαφορά στις απόψεις μου με τις απόψεις του κυρίου Οχτή για τα ευάλωτα άτομα, σε κάθε περίπτωση οι νομικοί που στελεχώνουν το Διαιτητικό Δικαστήριο είναι πολύ αξιόλογοι, ασχολούνται με το γενικότερο συμφέρον περισσότερο και πολύ λιγότερο με το να κάνουν πολιτική και αυτό μας καθησυχάζει. Είναι πολύ καλό. Επίσης είδα το πίνακα, το, την, το νεαρό κορίτσι με το σκουλαρίκι του Φερμίερ, του ζωγράφου. Είχα αυτή την ευκαιρία και έτσι συνειδητοποίησα ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί στην Ευρώπη, αλλά έχουμε κοινούς στόχους, κοινά ιδεώδη, κοινό πολιτισμό και αξίζει τον κόπο να τον υπερασπιστούμε. Αυτός είναι ο απολογισμός της μου και από όλε τι αποστολέ στις οποίε έχω συμμετάσχει αυτή ήταν και η πιο ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε πολύ ε, αναζωογονητικά αυτά που μα είπατε. Κυρία Ρέντα, θέλετε να μα σχολιάσετε και εσεί την αποστολή στην Ουτρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για μια πολύ καλά οργανωμένη αποστολή η οποία μας έδωσε μια λεπτομερή εικόνα των δραστηριοτήτων της Επιτροπής σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Δύο τομείς είναι αυτοί οι οποίοι μου φάνηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντες. Πρώτον, είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε μια συζήτηση πανεπιστημιακού επίπεδου για τις βασικές αρχές που διέπουν ακριβώς με τη σειρά τους την αρχή της της καλύτερης νομοθετικής δραστηριότητας, της βελτιστοποίησης της νομοθετικής παραγωγής. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται στην μεταφορά των πολιτικών ιδεών σε νομοθετικό επίπεδο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο πνεύμα αυτών που επιθυμούν οι πολιτικοί και να μην έχουν άμεσα ένα πολιτικό περιεχόμενο και όχι απλά μείωση του γραφειοκρατικού ε, βάρους. Έγινε μια συζήτηση λοιπόν ανάμεσα σε πανεπιστημιακούς και σε εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και είδα τις διαφορές αυτές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Επίσης επισκεφθήκαμε και μαζί μάλλον έγινε και επίσκεψη με το Eurojust Κάποιες από τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες ακολούθησαν τον Σεπτέμβριο την επίθεση την τρομοκρατική είναι κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να επανεξεταστούν να υπήρξε μια υπεραντίδραση σε πολιτικό επίπεδο και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και σε νομικό επίπεδο δεν ήταν τα καλύτερα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία ήταν ο βασικός στόχος. Έγιναν επίσης και συζητήσεις για κάποια άλλα θέματα όπως τα θέματα του Διοικητικού Συμβούλου Επιχειρήσεων είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε εμείς την προσπάθειά μας. Ήταν πολλά εμπασπέρτος τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Έγιναν επίσης και κάποιες περαιτέρω συζητήσεις ε, για, τα, για τις πιθανότητες δημιουργίας των διεθνών ιδιωτικών διαιτητικών δικαστηρίων. Θα πρέπει να πάρουμε μια πολιτική απόφαση αν θέλουμε να προστατεύσουμε με τέτοιο τρόπο τις επενδύσεις ε, στην περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση με τα δημόσιο συμφέρον και μετά να δούμε πώς θα οργανωθεί ένα τέτοιο ε, διαιτητικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άουταλα. Και εγώ νομίζω ότι άξιζαν αυτές οι δύο ημέρες. Υπήρξαν πάρα πολλές συναντήσεις. Υπήρξε μια σαφής κατανόηση της λειτουργίας, σε βάση περιπτώσει, των διεθνών οργανισμών σε επίπεδο διεθνούς δικαίου στη Χάγη. Είχαμε μια πολύ θερμή συνάντηση με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, την Επιτροπή για το Ιδιωτικό Διεθνές της Χάγης. Είναι κεντρική αρμοδιότητα της Επιτροπή μας και θεώρησαν ότι η επίσκεψη ήταν σημαντική και για αυτούς, όχι μόνο για μας. Θα πρέπει να είμαστε σε στενή επαφή μαζί τους να συνεχίσουμε τις συζητήσεις ε, για θέματα δύσκολα. όπως το πώς μπορούμε σε διεθνές επίπεδο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα κληρονομίας κτλ. Μία από τις εκπλήξεις της επίσκεψης αυτής είναι ότι κανένα κοινοβουλευτικό σώμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε επισκεφθεί το μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο και αυτό ήταν έκπληξη για μας και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η κυρία Ρέντα. Είναι ένα σημαντικό θέμα το θέμα της διαιτησίας. Πρώτα θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι τα επίπεδα δημοσίου συμφέροντος τα οποία θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο προστασίας πριν πάρουμε αποφάσεις για διαιτητικά. Και το Eurojust είναι ένας θεσμός που δεν χρησιμοποιείται πλήρως νομίζω αλλά η εμπλοκή τους στην αναζήτηση ή στις ανακρίσεις και στις διώξεις μάλλον σε επίπεδο ε, καταπολέμησης ε, της διεθνούς εγκληματικότητας είναι χρήσιμη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να εξετάσουμε εγκύτερα τις ανάγκες ε, της Eurojust. Από ό,τι φαίνεται επίσης πρόκειται για ένα θεσμό ο οποίος είναι υποχρηματοδοτούμενος και αυτός και να προσθέσω μία επιπλέον παρατήρηση σε ένα από τα προηγούμενα θέματα σήμερα θέσαμε το θέμα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στις χώρες με εταιρική σχέση, με διαδικασία ένταξης έχουν υποτίθεται μια συμφωνία και με τη Eurojust. Σαν παράδειγμα όταν δημιουργείται μια κατάσταση όπως η σημερινή στη Μολδαβία όπου υπάρχει μια κατάχρηση μεγάλου μεγέθους στην κεντρική τράπεζα και σε άλλες τράπεζες θα πρέπει η Eurojust να ενημερώνεται για τις έρευνες. Λοιπόν, πάντως νομίζω ότι ήταν μια καλή αποστολή και δεν ήταν σε μια μακρινή χώρα δεν κράτησε πολλές μέρες, αλλά έχω μια πολύ καλή εντύπωση για το πώς εργάζονται οι θεσμοί της Χάγης. Ήταν σημαντικό ότι είχαμε μια ιδιωτική συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ολλανδίας που έχει έρθει εδώ στην Επιτροπή και κάναμε συζητήσεις που είχαμε ξανακάνει στο παρελθόν μαζί του σε τομείς όπου η Ιλλανδική Προεδρία θέλει να προχωρήσει και να χρησιμοποιήσει επίσης και ε, για ειδικά καθεστώτα γάμου και ε, περιουσιακές σχέσεις των συζύγων την ενισχυμένη συνεργασία. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας και την ενημέρωση από την αποστολή αυτή. Κάνατε μία παρατήρηση κυρία Χάουταλα σχετικά με τις εξωτερικές υπηρεσίες. Μιλήσατε για το Eurojust που έχει ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό. Είναι βασικό πρόβλημα των οργάνων μας να δημιουργούμε εξωτερικές υπηρεσίες και να τις πρικίζουμε με ελάχιστα χρήματα. Ξέρουμε το Frontex το οποίο έχει αναλάβει τρομακτικές ευθύνες ενώ του μειώνουμε συστηματικά τα οικονομικά μέσα για να φέρει εις πέρας την αποστολή την οποία του έχουμε αναθέσει. Ακούσαμε λοιπόν τις ευχαριστίες των συναδέλφων ε, αν πεθύνομαι στα μέλη της γραμματείας και σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στο 12 και 13 για τον συνάδελφο Λεμπρετό. Ευχαριστώ <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Για το 12 είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2008-98 για τα απόβλητα. Είναι ένα πακέτο με τις τροποποιήσεις οδηγιών στα σημεία 14, 15 και 16. Όλες για τα απόβλητα. Το πλαίσιο της πρότασης είναι το εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει ένα τεράστιο ποσό πρώτων υλών μέσω της απώλειας των αποβλήτων. Η παραγωγή αποβλήτων είναι πάνω από δις τόνους και ένα δις 600 εκατομμύρια χάθηκαν χωρίς ανακύκλωση. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η χρήση των πόρων από τα απόβλητα και να ενισχυθεί η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Εκεί είναι το βασικό στόχος. Οι εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις δεν είναι ομοιογενείς για τη διαχείριση των αποβλήτων. Το 2011 μόνο το 3% των δημοτικών αποβλήτων έθεταν σε, σε ανακύκλωση ένα 6-7% ενώ άλλες χώρες ξεπερνούσαν το 50%. Αυτές οι τέσσερις λοιπόν οδηγίες, οι, μετα... οι τροποποιήσεις των οδηγιών έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Τίθεται εδώ το θέμα της αρχής της επικουρικότητας, επί της οποίας πρέπει να εκφραστούμε. Δύο εθνικά κοινοβούλια έχουν εκφέρει τεκμηριωμένες συστάσεις. Η Γαλλική Γερουσία στις 2 Φεβρουαρίου του 2016 και το Ανώτατο Συνταγματικό Αυστριακό Συμβούλιο θεωρούν ότι η πρόταση οδηγίας δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας. Εγώ νομίζω ότι έχουν δίκιο, πρέπει να σας πω και εγώ την άποψή μου και θα σας ε, παρουσιάσω έξι επιχειρήματα για να προσπαθήσω να σας πείσω είναι επιχειρήματα τα οποία περιλαμβάνονται και στα έγγραφα των δύο αυτών κοινοβουλευτικών οργάνων. Πρώτο επιχείρημα από το Ομοσπονδιακό Αυστριακό Συμβούλιο. Οι Αυστριακοί θεωρούν ότι στην οδηγία αυτή υπάρχει μια ατελής ε, προσπάθεια ορισμού του τι είναι δημοτικό ή κοινοτικό απόβλητο. Ε, λαμβάνονται υπόψη αυστηρά ποσοτικά κριτήρια, γιατί τα απόβλητα αυτά δεν θεωρούνται δημοτικά παρά μόνο πάνω από ένα όγκο. Κάτι το οποίο είναι περίεργο και ανησυχεί το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Η ίδια τεκμηρίωση αφορά επίσης ε, και τα λεγόμενα βιοαπόβλητα και τον ορισμό των βιοαπόβλητων. Βασίζεται σε αποκλειστικά ποσοτικές μεθόδους Δεύτερο επιχείρημα εναντίον της συγκεκριμένης πρότασης αλλαγής της οδηγίας και είναι το μείζον επιχείρημα της γαλλικής γερουσίας. Κάθε φορά υπάρχει μια ε, ευρυτάτη προσφυγή στις εκτελεστικές πράξεις και στις κατεξουσιοδότηση πράξεις, όχι για μικρές λεπτομέρειες αλλά για οσιώδη θέματα ο καθορισμός των δικτών επιδόσεων σε σχέση με την πρόληψη ε, της, ε, των αποβλήτων για τα ποσοτικά ε, όρια, τα ανώτητα μη επικίνδυνων αποβλήτων ή επίσης και για τον καθορισμό των επίσημων δικτύων συλλογής. Λοιπόν, ε, εγώ δεν σας παραπέμπω στον τεράστιο αριθμό των άρθρων, αλλά είναι εντυπωσιακά τα επιχειρήματα αυτά. Η Γαλλική Γερουσία λοιπόν πιστεύει ότι αυτή η μαζική προσφυγή σε εκτελεστικές πράξεις και κατεξουσιοδότηση πράξης παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει να πω ότι ο φόβος αυτός έχει ήδη διατυπωθεί εδώ και κάποια χρόνια από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Γερουσίας. Είναι η έκθεση Σιμών Σιτούρ του 14, Φεβρουάριο του 14. Και γι' αυτό η ειδική αυτή επιτροπή καταδικάζει αυτή την τάση πολλαπλασιασμού των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Ίσως είναι λοιπόν ένας τρόπος διακριτικής παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας. Δεν πρόκειται για μια ξεκάθαρη παραβίαση μέσω της οδηγίας, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται με έμεσο τρόπο από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Δεν το λέω εγώ, το λέει η έκθεση Σιμό Σιτούρ. Ο γερουσιαστής αυτής, ή μάλλον οι γερουσιαστές αυτοί πήραν μέρος στη συζήτηση που έγινε και στην πρώτη συζήτηση ήδη από το 2007. Τρίτο επιχείρημα το άρθρο 9 της πρότασης οδηγίας την οποία συζητάμε σήμερα επιβάλλει στα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο διαμαρτύρεται γιατί θεωρεί ότι αυτή η υποχρέωση περιορίζει τις δυνατότητες δράσης των κρατών μελών πιστεύουν ότι η αρχή της επικουρικότητας στα πλαίσια του μέτρου αυτού αλλοιώνεται επειδή καλούμεθα να πάρουμε μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, κάτι το οποίο δίδει υπερβολικές εξουσίες ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέταρτο επιχείρημα, ανακοίνωση της ε, ετήσιας και σαν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό θα δημιουργήσει ε, διαδικασίες γραφειοκρατικές ιδιαίτερα βεβαρημένες και τα επεξηγηματικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν τις αποφάσεις αυτές θα είναι δύσκολο να συνταχθούν όπως και οι πίνακες ταύτισης οι οποίοι θα πρέπει να διευκρινίζουν ποιο είναι το τμήμα της οδηγίας που μετετέθη και εφαρμόστηκε σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας. Ε, επιπλέον γραφειοκρατικά βάρη τα οποία δεν σέβονται κατά τη γνώμη των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων την επικουρικότητα. Πέμπτο επιχείρημα. Η Γαλλική Γερουσία καταδικάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τους όρους αξιοποίηση και εξαφάνιση των αποβλήτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει κάποιες εθνικές πρακτικές οι οποίες μπορούν να λάβουν υπόψη καλύτερα τις τοπικές συνθήκες αποβλήτων. Έκτο τελικά επιχείρημα, οι Γάλλοι γερουσιαστές θεωρούν ότι η έκθεση προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση ε, παραβάσεως ε, ή μη ανάληψης δράσης από τα κράτη-μέλη είναι υπερβολικά δεσμευτικό. Παράδειγμα, ε, οικονομικά κίνητρα προβλέπονται ενώ τα θέματα φορολογίας σαν παράδειγμα άπτονται αυστηρά της πολιτικής των κρατών μελών. Και εδώ η μη ανάληψη δρασης απο τα κρατη μελη ειναι υπερβολικα δεσμευτικο παραδειγμα οικονομικα κινητρα προβλεπονται ενω τα θεματα φορολογιας σαν παραδειγμα απτονται αυστηρα της επικουρικότητας δεν γίνεται σεβαστή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία λέγουν οι Αυστριακοί και οι Γάλλοι και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πακέτο για τα απόβλητα παραγνωρίζει επανειλημμένα έξι φορές την αρχή της επικουρικότητας. κύριος Καβαντά θέλει το λόγο. Να δείξω τι εννοεί ο κύριος Λεμπρετό στην περίπτωση που γνωρίζω τη γαλλική γερουσία εννοώ. Η έκθεση Σίμων Σιτούρ δεν είναι η έκθεση ενός παρανοϊκού αντιευρωπαίου, γιατί ήταν μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και γι' αυτό τα επιχειρήματά του θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ο κύριος Μαρίνιο Επίντου. Σε σχέση με αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι ε, η επικουρικότητα είναι το σχετικό και θέλω να αναφερθώ στο θέμα των απορριμμάτων και των αποβλήτων γενικότερα. Στην κοινωνία της κατανάλωσης, στην εκβιομηχανισμένη κοινωνία της κατανάλωσης και φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία οργανώτα, οργανώνεται γύρω από το τοτέμε της ανάπτυξης. Είναι ο Θεός μας. Θα πρέπει κάθε χρόνο να υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό είναι μια σταθερά. Και αναρωτιέμαι, τι ερωτήσεις. Είναι, μπορεί αυτός πραγματικά να είναι πολιτικός σκοπός, να είναι στόχος σε ένα πλανήτη τον, του οποίου οι πόροι είναι πεπερασμένοι. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να αναπτύσσεται δεν θα υπάρχει άλλος χώρος για ανάπτυξη ή εν περιπτώσει ο όρος ανάπτυξη πρέπει να αλλάξει περιεχόμενο και νόημα. Θα έρθει κάποια στιγμή όπου θα πρέπει να καταναλώσουμε λιγότερο ή κάποιοι τέλος πάντων να καταναλώσουν λιγότερα έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να καταναλώσουν καλύτερα, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα. Και τα απορρίμματα και τα απόβλητα, είτε οικιακά είτε βιομηχανικά, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης με διαφορετική οπτική γωνία. Τα οικιακά απορρίμματα οφείλονται κυρίως στην κοινωνία της κατανάλωσης. Υπάρχει αδιφαγία, υπάρχει μία αιμονή στα ψώνια και στις αγορές. Αγοράζουμε, καταναλώνουμε, αγοράζουμε, εξοδεύουμε, καταναλώνουμε, αγοράζουμε, εξοδεύουμε, καταναλώνουμε. Αυτό είναι καλό για την απασχόληση ενδεχομένως ή την οικονομία και, και έχει γίνει πια, ε, έχει μυθοποιηθεί θα έλεγα. Επομένως, οικιακά απορρίμματα θα μειώσουμε, μειώνοντας, έχοντας μια πιο σόφρονα κατανάλωση. Έχουμε τώρα και τα βιομηχανικά απορρίμματα και απόβλητα. Έχουμε, για παράδειγμα, τα πυρηνικά απόβλητα. Εκεί ε, οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε ότι για να ανακυκλωθούν θα χρειαστούν χιλιάδες χρόνια. Η ανακύκλωση είναι πολύ πιο εύκολη για τα οικιακά απορρίμματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλο μέρος της παραγωγής ενέργειας, ε, ε, ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με ε, την πυρηνική. Τι θα κάνουμε λοιπόν με τα απόβλητα αυτής. Πώς θα τα επεξεργαστούμε. Γίνεται λόγος ε, για την αποστολή όλων αυτών των αποβλήτων στο διάστημα, σε άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Νομίζω ότι η πρόταση αυτής της οδηγίας για την επικράτηση της αρχής της επικουρικότητας ε, θα πρέπει να υπερισχύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή επεξεργασία οικιακών απορριμμάτων και αποβλήτων, έτσι ώστε η βιομηχανία να έχει πηγή ενέργειας τα απορρίμματα και τα απόβλητα. Υπάρχουν εφαρμογές και στο επίπεδο της πυρηνικής ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, όλα αυτά δεν συνδέονται με την επικουρικότητα. Ο κύριος Πίντο. Όχι, δεν συνδέονται με την επικουρικότητα. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που έκανα, ή μάλλον ναι, σημείο εκκίνησης είναι η επικουρικότητα. Όμως προσπάθησα επί της ουσίας να θίξω το θέμα, να τοποθετηθώ πολιτικά. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει κεντρικά να διαχειριστεί το θέμα των απορριμμάτων και των αποβλήτων και των καταλήπων να είναι ένας ε, στόχος αυτός μέσω μακροπρόθεσμος. Επιμένω στο γεγονός ότι ε, σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να επιβάλλει πολιτικές εξαιρετικά θετικές στα κράτη-μέλη. Στην Πορτογαλία για παράδειγμα, όπου δεν υπήρχε καθόλου η νοοτροπία του σεβασμού στο περιβάλλον. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώσαμε αυτές τις πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε την πολιτική αυτή στην Πορτογαλία προς όφελος του πορτογαλικού λαού. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διακόψουμε μέχρι τις 11.30 διότι τότε θα έρθει ο Αντώνιο Καμπίνιο, πρόεδρος του Γραφείου για την Αναρμόνιση στην Εσωτερική Αγορά. Κύριε Λεμπρετό, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Ναι. Κοιτάξτε, Μίλησα μόνο για τα απορρίμματα και τα απόβλητα, αλλά υπάρχει και το 13 για τα όπλα. Ο πρόεδρος. Είχα κατανοήσει, είχα καταλάβει ότι όλα τα ε, σχολιάζεται συνολικά. Όχι, όχι, λέει ο κύριος Λεμπρέτον. Όχι, τα όπλα δεν έχουν καμία σχέση με τα απόβλητα και τα απορρίμματα, κύριε Πρόεδρε. Επομένως δεν έθιξα καθόλου αυτό το θέμα. Μου δίνετε τώρα το δικαίωμα να το κάνω. Σημείο 13 έλεγχος της κτήσης και κατοχής των όπλων. Ε, αφορμή και αφετηρία ήταν τα θλιβερά γεγονότα του Παρισιού του Νοεμβρίου της περασμένης χρονιάς. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι για την κτήση και την αγορά και την κατοχή των όπλων. Πολλαπλή είναι η στόχη αυτού του κειμένου. Πιο αυστηροί κανόνες για την ε, κράτηση, ε, κατοχή ορισμένων ή μη αυτόματων πυροβόλων όπλων. Πιο αυστηρές προϋποθέσεις για τη διαδικτυακή αγορά πυροβόλων όπλων. Κοινή οι κανόνες για την ετικετοθεσία, τη σήμανση των όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε καλύτερη ανιχνευσιμότητα ή χνηλασιμότητα αυτών, βελτίωση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, διασύνδεση των εθνικών μητρώων κατόχων όπλων και θέλουμε να παρεμποδίσουμε την μετατροπή σε πραγματικά πυροβολά όπλα ε, διαφόρων εξαρτημάτων και εργαλείων και ενίσχυση των προϋποθέσεων και συνθήκων που πρέπει να τηρούν οι συλλέκτες, για, συλλέκτες όπλων για να μειωθεί ο κίνδυνος να μεταπουλήσουν αυτά τα όπλα ε, τα συλλεκτικά σε τρομοκράτες. Πολύ φιλόδοξη όλη αυτή η στόχη βασική βάση είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα επιτρέπεται η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών έτσι ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά. Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική, κυρίως ως προς το κατά πόσο τηρείται ή όχι η αρχή της επικουρικότητας. Νομική κριτική δηλαδή. Δύο αιτιολογημένες γνώμες λάβαμε, μία από το Σουηδικό Κοινοβούλιο εξαιρετικά ενδελεχή και μία άλλη εξαιρετικά ρίζοσπαστική από την Πολωνική Γερουσία. Θα σχολιάσω αυτές τις γνωμοδοτήσεις και κυρίως την άποψη του Σουηδικού Κοινοβουλίου για να σας εξηγήσω ότι κατά τη γνώμη μου η πρόταση αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα και έχω θα απαριθμίσω 7. Πρώτο πρόβλημα είναι δύσκολο να ξέρει κανείς σε ποιο βαθμό ο περιορισμός της διάρκειας ισχύω των αδειών και των υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων του κατόχου του όπλου πράγματι θα αυξήσει την ασφάλεια του πολίτη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέται κανείς αν αυτή η πρόταση του περιορισμού της χρονικής διάρκειας της ισχύω της άδεια δεν ε, ε, ε, υπονομεύει την αρχή της επικουρικότητας. Δεύτερο, πρόταση να συμπεριληφθούν τα όπλα που εκτίθενται στα μουσεία είναι υπερβολικό για το Σουηδικό Κοινοβούλιο, διότι είναι μάλλον απίθανο <laughs> τέτοια όπλα να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, στο βαθμό που τα μουσεία, εν περιπτώσει, έχουν κανόνες ασφαλείας αρκετά σημαντικούς. Τρίτον, η πρόταση θέλει να περιορίσει το εμπόριο των όπλων μεταξύ ιδιωτών, όμως πάει πάρα πολύ μακριά. Ε, θεωρεί το Σουηδικό Κοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια πιο λεπτομερή επιχειρηματολογία ως προς το γιατί και το πόσο περιορισμός και ο έλεγχος του εμπορίου μεταξύ ιδιωτών είναι απαραίτητος για την καταπολέμηση της, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το Κοινοβούλιο λοιπόν, το Σουηδικό δικαίω κατά την άποψή μου ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αιτιολογήσει περισσότερο τις προτάσεις της. Τέταρτο πρόβλημα, ορισμένα μέρη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ασαφή, ορισμένα τμήματα και περιπλέκουν την αξιολόγηση για το κατά πόσο εφαρμόζεται η επικουρικότητα. Μιλούμε για πυροβόλα όπλα τα οποία φαινομενικά φαίνονται αυτόματα, αλλά δεν είναι αυτόματα όπλα. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς και ποια είναι αυτή η κατηγορία των όπλων. Άλλωστε πολλές διαμαρτυρίες και πολλά προβλήματα δημιουργούνται με αυτή την περιγραφή, την ασαφή και την ατελή περιγραφή. Τώρα, πέμπτο πρόβλημα και συμφωνεί με αυτό η πολωνική γερουσία. Τα επιχειρήματα στο αιτιολογικό δεν καταδνύουν ότι ο περιορισμός του υπεριορισμού που επιβάλλονται στο εμπόριο όπλων μεταξύ ιδιωτών θα συμβάλλουν πραγματικά στη μείωση της τρομοκρατίας. Ότι υπάρχουν δηλαδή άλλα μέτρα πολύ πιο αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το αγαπημένο μου από αυτά είναι βεβαίως η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Έτσι καταπολεμάται η τρομοκρατία και όχι με τους περιορισμούς τους αυστηρούς στο εμπόριο μεταξύ ιδιωτών. Τώρα, έκτον, ε, γίνεται αναφορά σε αρνητικές συνέπειες προβλεπόμενες. Το, η αγορά του εμπορίου όπλων θα είναι πολύ πιο δύσκολη, ε, θα υπάρξει επίπτωση στις θέσεις απασχόλησης και θα χάσουν την αξία τους οι συλλογές. Γιατί αφού θα πρέπει να είναι αποενεργοποιημένα τα όπλα που είναι συλλεκτικά, τότε η συλλογή χάνει την αξία της την εμπορική, την οικονομική. Θα υπάρξει διοικητικό κόστος και θα πρέπει να υπάρξει αποσμίωση των ιδιοκτών, ε, με την κατάσχεση βεβαίως ορισμένων όπλων. Θα δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα εκεί σε αυτό το επίπεδο. Έβδομο επιχείρημα. Οι περιορισμοί που προτείνονται για την όμιμη κατοχή πυροβόλων όπλων σύμφωνα με την Πολωνική Γερουσία αλλά και το Σουηδικό Κοινοβούλιο επιβάλλουν αδικαιολόγητους περιορισμούς σε τρεις κατηγορίες χρηστών τους κυνηγού, όσοι είναι σκοπευτές για λόγους άθλησης και ψυχαγωγικούς και τους συλλέκτες. Πλήτεται το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην ιδιοκτησία, στην περιουσία και βεβαίως δεν μπορούν ελευθέρως να χρησιμοποιήσουν ε, τα αγαθά των οποίων είναι ιδιοκτήτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόλου δεν αποδεικνύει ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι κατάλληλοι και ταιριάζουν με τον υποτίθεται στόχο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της πολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων. Καθόλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το αποδεικνύει αυτό. Και όταν η Επιτροπή λέει ότι τίποτα δεν θα αλλάξει για τους κυνηγού και για τους ε, αθλητικούς ε, σκοπευτές, όσοι ασχολούνται με τη σκοποβολή για λόγους ψυχαγωγίας και αθλητικού. Ε, δεν το αποδεικνύει. Σίγουρα θα υπάρχουν νομικές συνέπειες για τους νόμιμους χρήστες ε, των όπλων, οι οποίοι βεβαίως και τηρούν την νομοθεσία. Κάτι πολύ συγκεκριμένο που ενοχλεί ιδιαιτέρως τους ε, κυνηγούς και τους σκοπευτές είναι η πρόταση απαγόρευσης των ημιαυτόματων όπλων που τώρα εντάσσονται στην κατηγορία Β7 και χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους κυνηγού αλλά και από τους αθλητές του αθλήματος της κοποβολής. Είναι υπερβολική αυτή η απαγόρευση σε σχέση με τον ε, ε, στόχο. Και για να συνοψίσω, αυτή η οδηγία δεν επιλύει κανένα πρόβλημα ε, ως προς την παράνομη κυκλοφορία παρανόμων ε, όπλων. Ε, αντίθετα, δημιουργεί επιπρόσθετα βάρη για τους πολίτες που χρησιμοποιούν τα όπλα νομίμως. Και δεν επιτυχάνει τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι δυσανάλογοι οι περιορισμοί που επιβάλλονται και παρακάμπτεται η αρχή της επικουρικότητας και Οπότε το συμπέρασμά μου είναι ότι κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ε, δημιούργησε μεγάλη πόλωση στράφηκε εναντίον των πυροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται νομίμως, ενώ οι τρομοκράτες δεν έχουν αυτά τα όπλα στη φαρέτρα τους, αντιθέτως εξοπλίζονται με όπλα που κυκλοφορούν στο λαθρεμπόριο. Η Επιτροπή λοιπόν θυσιάζει τα ε, νόμιμα εμπορικώς ε, ε, χρησιμοποιούμενα όπλα για να πετύχει το στόχο της και δεν τον καταφέρνει ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρίνιο Πίντο. Ευχαριστώ. Όπως και στο προηγούμενο θέμα, θέλω να πω για την επικουρικότητα, αλλά γενικά για τα όπλα, καταρχήν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει πιο σκληρά απαγορευτικά μέτρα. Να είναι αδύνατον να πολιθεί όπλο, για παράδειγμα, αν ένα πολίτη δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπως εγώ δεν μπορώ. Το ότι όλοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αυτό είναι κίνδυνος. Ο κόσμος θα ήταν πολύ ασφαλέστερος και πιο ειρηνικός αν μπορούσαμε να απο... απαγορεύσουμε τελείως τη χρήση όπλων. Ο κόσμος... Ε, ίσως να ακούγεται αυτό σαν γλάστος για ορισμένους, αλλά αν μπορούσαμε να απαγορεύσουμε το κυνήγι κάποιων ειδών θα ήταν καλό γιατί δεν είναι, δεν είναι ε, αθλητική δραστηριότητα να σκοτώνεις τα πουλιά ή να ε, βασανίζεις τα ζώα. Προέρχομαι από χωρο που δεκάδες είδη πουλιών έρχονται την Άνοιξη στην Πορτογαλία και κάποια είδη κάνουν τη φωλιά τους την εποχή που αρχίζει η εποχή του κυνηγιού για να τα πυροβολούν και να τα σκοτώνουν. Αυτό είναι α, ε, ε, ε, απαράδεκτη αγριότητα. Πάντα είναι λάθος να σκοτώνει ζωντανά πλάσματα. Δεν είναι αθλητισμός αυτός. Δεν είναι σωστό να το επιτρέπεις, γιατί η ιδέα του αθλητισμού δεν πρέπει να συνεπάγεται θανάτωση ποτέ. Ξέρω ότι υπάρχουν παλιοί μύθοι και στη Βραζιλία έγινε ε, δημοψήφισμα πρόσφατα για να απαγορευτεί το εμπόριο ε, όπλων για άμυνα. Και το, ο αντίλογος ήταν ότι μόνο οι ληστές θα ήταν οπλισμένοι για αυτή την περίπτωση. Πάντως, ένας μακροπρόθεσμος στόχος όλο τον κόσμο πρέπει να είναι η απαγόρευση της χρήσης των όπλων. Η ασφάλεια των ανθρώπων δεν ε, ενισχύεται με την κατοχή όπλων. Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια μέσα από τους κανόνες κοινωνικής συμβίωσης και μέσα από τον νόμο και την τάξη και τις αστυνομικές αρχές. Εκείνοι να έχουν τα όπλα. Εκείνοι μόνο πρέπει να έχουν και η χρήση των όπλων μάλιστα από τις αστυνομικές αρχές επίσης θα πρέπει να είναι σαφώς προδιαγεγραμμένη. οι τρομοκράτε δεν πηγαίνουν σε κανονικά οπλοπολία να αγοράσουν. Είναι διαφορετικό το θέμα. Εκείνοι κινούνται στην παρανομία. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε σε πολιτικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να ελέγξουμε την ε, βιομηχανία όπλων και να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια εκεί. Γιατί βέβαια η συμβολή στο ΑΕΠ πολλών χωρών, το, Κίνας, ΙΠΑ, ε, βέβαια αυτό υπάρχει. Ε, κάνουν εξαγωγή όπλων κρυφά και παράνομα πολλές φορές τροφοδοτώντας περιφερειακές συγκρούσεις σε διαρκή βάση. Ε, δείτε σε κάποια μέρη της Αφρικής ε, που μάχονται μεταξύ τους οι φυλές. Πρέπει να είναι δυνατόν να τα βελτιώσουμε τα πράγματα, να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα. Κανείς καλοπροαίρετος άνθρωπος δεν χρειάζεται όπλο να το κατέχει. Μπορεί να ε, γίνει επίθεση, αλλά α, διακόπτει ο πρόεδρος. Και για την ε, επικουρικότητα, τι έχετε να πείτε. Ναι, ναι, μου φαίνεται παρασύρθηκα λιγάκι, συγγνώμη. Ξέχασα τη σύνδεση με την επικουρικότητα. Για να τελειώνω, γιατί έχουμε και πολλά ακόμα, ε, θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο χωρίς όπλα. Και παρασύρθηκα λίγο, γιατί ε, με τα όπλα. Ευχαριστώ, κυρία Χάουταλα. Η πρόταση της Κομισιόν προκάλεσε πολλές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σε πολλά κράτη-μέλη. Εν μέρη ε, ο λόγος υπάρχει στις νομοδοτήσεις για την επικουρικότητα από τα κοινοβούλια Πολωνίας και Σουηδίας. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε την πρόταση μέσα από το πρίσμα της επικουρικότητας. Οπότε δεν θα ήμουν υπέρ της επίκλησης ε, της επικουρικότητας. Όμως μπορούμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Φαίνεται ότι η πρόταση που είναι τώρα στα χέρια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς του Κοινοβουλίου με γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών και άλλες ίσως μπορεί να αναφερθούν σε κάποιες πτυχές της πρότασης που ίσως δεν χρειάζονται 100% πάντα έχοντας κατά το σκοπό της οδηγίας, της πρότασης. Ίσως το Κοινοβούλιο λοιπόν μπορεί να δει και το θέμα της ε, αναλογικότητας και αν έχει παραβιαστεί αυτό. Αυτό οι επιτροπές επί της ουσίας μπορούν να το κάνουν. Πάντως ε, αληθεύει ότι υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν την ε, εκτίμηση των επιπτώσεων, την συμπερίληψη κάποιων κατηγοριών όπλων πάντα έχοντας υπόψη το σκοπό της ε, πρότασης, δηλαδή που είναι η παροχή δημόσιας ασφάλειας ε, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά αυτό ίσως είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να επικαλεστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Ο κύριος Λεμπρετών να πει κάποια άλλα πράγματα. Να ευχαριστήσω τους κυρίους κυρίους Πίντο και Χάουταλα για τα σχόλια τους. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Χάουταλα ότι αυτή η πρόταση οδηγίας δημιουργεί θέματα και σε επίπεδο αναλογικότητας. Αυτό είναι αληθές. Και πρέπει να επανεξεταστεί η πρόταση αυτή η οποία δεν μου φαίνεται σωστή. Σχετικά με τις απόψεις του κυρίου Πίντο θέλω να τον διαβεβαιώσω. Εγώ είμαι υπέρ της χρήσης των ιδιωτικών όπλων δεν είναι για αυτό άμυνα. Δεν συμφωνούμε με τους Αμερικανούς ή Γάλλοι. Νομίζω ότι υπάρχουν νόμιμοι τρόποι χρήσης των όπλων. Αναφέρθηκα σε δύο. Καταρχάς η σκοποβολή είναι καταρχα η σκοποβολη ειναι κατι το οποίο εγώ δεν, ε, δεν κάνω, αλλά παρόλα αυτά είναι μια αθλητική δραστηριότητα. Γιατί να καταργηθεί μια αθώα τέτοια δραστηριότητα. Και η δεύτερη δραστηριότητα είναι το κυνήγι. Το κυνήγι δεν είναι πολύ κακό πράγμα κύριε Πίντο. Ήμουνα κυνηγό όταν ήμουν νέος. Και δεν είναι θέμα προσωπικής ευχαρίστησης, είναι δημόσια υπηρεσία στη Γαλλία. Είναι δραστηριότητα κοινή ωφέλεια, διότι στόχος είναι η συντήρηση της πανίδας. Όταν είναι σωστά οργανωμένη, ρυθμίζει τον πληθυσμό των ζώων και δεν το καταστρέφει και πρόσφατα ε, πήγαν αγριογούρουνα στο Φοντεμπλό γιατί είναι δυστυχώς πάρα πολλά. Αυτό λοιπόν επιτρέπει να το λύσουμε το κυνήγι. Σας ευχαριστώ. Αν η Επιτροπή της ΣΥΜΚΟ είχε όπλο θα μας πυροβολούσε γιατί τα θέματα αυτά είναι δικής της αρμοδιότητας. Λοιπόν, πέραν αυτού νομίζω ότι τώρα θα διακόψουμε μέχρι τις 11.30 για τον... Ε, για να υποδεχθούμε τον κύριο Καμπίνος. Ε, με έχει ο κύριος ε, Μαρίνιο Επίντο εδώ στην Επάρη. Ζητώ συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει το λόγο, γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι παρακαλώ να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λίγο. Έχει ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, σύντομα, Πρόεδρε, για το θέμα της επικουρικότητας. Είναι ένα πολύ σημαντικό φυσικά θέμα. Νομίζω ότι πράγματι εμείς ενημερωθήκαμε για την γνωμοδότηση ε, της Σουηδικής Βουλής και της Πολωνικής Βουλής και η Ιταλική Γερουσία εξεφράστηκε από αυτού και θεώρησε ότι δεν ετίθεται το θέμα επικουρικότητας όπως και η Πορτογαλική ε, Γερουσία που διαπίστωσε έλλειψη προβλήματος. Πρέπει να αναφερθούμε στο σύνολο λοιπόν. Τώρα το θέμα της αναλογικότητας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σύντομα να αναφερθώ σε δύο ή τρία σημεία. Στόχος μας δεν είναι να καταπολεμήσουμε μόνο την τρομοκρατία. Το πρόβλημα των όπλων δεν είναι μόνο συνδεδεμένο με την τρομοκρατία. Πριν λίγα χρόνια εσφάγισαν 77 νέοι σε μία κατασκήνωση. Δεν είναι θέμα τρομοκρατίας ήταν ένας αθλητής σκοποβολής με νόμιμο όπλο που προκάλεσε αυτή τη σφαγή. Υπήρξαν σφαγές και σε σχολεία όπως το Όντεσεν στο Παρίσι και υπάρχουν μονίμως τέτοιου είδους απαράδεκτες ενέργειες με ημιαυτόματα πυροβόλα. Η μεγάλη πλειοψηφία βέβαια των συλλεκτών, των κυνηγών και των αθλητών δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Αυτό το αναγνωρίζουμε και να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα σύστημα που να μην επιτρέπει κατακρίσεις. Για τις τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι δεν είναι αλήθεια ότι τα όπλα είχαν έρθει από τη Συρία ή την Ανατολική Ευρώπη. Ένας από τους τρομοκράτες είχε ένα όπως λέγεται ακουστικό πυροβόλο ε, το αγοράζει κανείς ελεύθερα στην αγορά και με μια μικρή τροποποίηση μπορεί να χρησιμοποιείται για φόνους. Η κατηγορία P7 δεν είναι σαφής και πρέπει να το διευκρινίσουμε. Σε αυτή την κατηγορία Β7 περιλαμβάνονται επίσης τα καλάσνικοφ σαν παράδειγμα, τα οποία είναι ημιαυτόματα όπλα μεν, αλλά είναι καλάσνικοφ και ανάμεσα σε ένα αυτόματο και σε αυτόματο καλάσνικοφ αρκεί ένας μικρός διακόπτης για να αλλάξει η λειτουργία του όπλου. Στον Πατακλάνα είχαν αυτόματα Καλάσνικοφ αλλά χρησιμοποίησαν τα αυτόματα γιατί είναι πιο αποτελεσματικά, δεν μ' αρέσει το επίθετο, αλλά είναι πιο φωνικά σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα κινηματογράφο γιατί έτσι χάνει κανείς λιγότερες σφαίρες. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους της ΣΥΝΚΟ, θέλουμε να βελτιωθεί η πρόταση οδηγίας, αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο ασφαλείας η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τεκμηριωμένη. Αν κάποιες πλευρές είναι υπερβολικές να την βελτιώσουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα στον τομέα της ασφάλειας. Ευχαριστώ για αυτή τη σημαντική παρατήρηση. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Η τρίτη μου προσπάθεια λοιπόν να κάνουμε διάλειμμα επιτυγχάνει μέχρι τις 11.30. Dear uh, I think we Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντώνιο Καμπίνους, πρόεδρος του Κέντρου εναρμόνισης των μέτρων της εσωτερικής αγοράς μέχρι τις 31 Μαρτίου. Γιατί τότε θα αλλάξει όνομα η υπηρεσία αυτή. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι ο εξής. Ο κύριος Καμπίνιους θα μας παρουσιάσει το πολιετές πρόγραμμα στρατηγικής της υπηρεσίας του. Ο λόγος για τον οποίο θα το κάνει αυτό είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας πριν υιοθετήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να συζητηθεί και στη δική μας Επιτροπή. Χωρίς λοιπόν καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον κύριο Καμπίνος. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τους άλλους συναδέλφους ε, της ε, συγκεκριμένης υπηρεσίας. Έχετε το λόγο κύριε Καμπίνος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την τελευταία φορά που ήρθα στην Επιτροπή είχα ετοιμάσει μια ομιλία 20-25 λεπτά, μετά μου έδωσε 10 λεπτά ο Πρόεδρος, οπότε έπρεπε, έπρεπε να μην διαβάσω το λόγο μου. Οπότε τώρα κάποιες παρατηρήσεις θα κάνω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που είναι παραπάνω από πρόσκληση. Είναι εξάντε ε, ε, πρόσκληση με την έννοια ότι στις 23 Μαρτίου θα τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις μαζί με αλλαγές σημαντικές στους κανονισμούς. Η Κομισιόν τους υπέβαλε και το Κοινοβούλιο που ενέκρινε προβλέπει αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή θα έχει δύο ψήφους στο Διοικητικό Οικομισιόν και το Κοινοβούλιο μία. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο εκτελεστικός διευθυντής από πρόεδρος θα είμαι εκτελεστικός διευθυντής, διατηρώντας όμως το όνομά μου Αντώνιο Καμπίνιος, ο εκτελεστικός διευθυντής θα μπορεί να επεκτείνει ε, το όραμά του πριν αρχίσει την εντολή του και ε, το πολιετές πρόγραμμα εργασίας, το πολιετές στρατηγικό πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο πριν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για την Επιτροπή την ε, Προϋπολογισμού του Οργανισμού. Οπότε όπως σας είπα, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 23 Μαρτίου, ε, αλλά και πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, πιστεύουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλό είναι να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει απόψεις για τον οργανισμό την επόμενη πενταετία, γιατί το στρατηγικό πρόγραμμα καλύπτει την επόμενη πενταετία. Οπότε ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη σκληρή δουλειά που κάνατε για να ε, εγκριθεί ο κανονισμός. Όλοι θα λάβατε και ελπίζω να είχατε χρόνο να διαβάσατε το στρατηγικό πρόγραμμα του οργανισμού, η UIPO, δηλαδή του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ένωσης, και μπορέσατε να διαβάσετε το πρώτο αυτό σχέδιο που ετοιμάστηκε πάνω στη βάση ευρειών διαβουλεύσεων που άρχισαν στο τέλος του 2014 γιατί τότε θεωρούσαμε ότι θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός το 2015 οπότε δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φροντίσουμε να είναι όλα έτοιμα ε, για να υποβληθούν στο διοικητικό το 2015. Υπήρξαν καθυστερήσεις και καθυστερήσαμε το στρατηγικό πρόγραμμα για να αρχίσει όταν ολοκληρωθούν οι επίσημες διαβουλεύσεις. Έχουμε το προσωπικό μας, όλα τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποφανθούν. Ακούσαμε και τις ενώσεις, τις ιδιωτικές ενώσεις και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ε, τους μεγάλους ε, διεθνείς εταίρους μας, το EPO και ε, εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε τις απόψεις τους και καταλήξαμε στο πρώτο σχέδιο. Η διαδικασία διαβούλευση συνεχίζεται. Ε, προβλέπονται επίσημα οι διαβουλεύσεις. Ε, η Κομισιόν πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία. Οι υπηρεσίες διαβουλεύονται. Μέχρι τις 22 Μαρτίου έχουν προθεσμία για να υποβάλουν απόψεις επί του σχεδίου και θα συλλεγούν όλες αυτές οι απόψεις και θα υποβληθούν τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου στο Διοικητικό, Συμβούλιο για να αποφανθεί. Τι είναι αυτό το στρατηγικό πρόγραμμα όμως. Ε, είναι δυναμικό, εξελισσόμενο εξέλιξη, περί εξέλιξης πρόκειται παρά για επανάσταση. Βέβαια δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος για να το αξιολογήσω ε, αν είχε επιτυχία το πρώτο, αλλά αντικειμενικά αν δείτε τον, τον αριθμό των έργων που άρχισαν και το ποσοστό ολοκλήρωσης όλων αυτών των έργων, αν δείτε ότι Έχουμε περιορισμένο προπολογισμό. Αν δούμε την ικανοποίηση των χρηστών, αν δούμε και την ικανοποίηση των, του προσωπικού εσωτερικά, βλέπουμε ότι πάντα υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης ε, στην ποιότητα, στην ε, εμπλοκή. Ε, είναι καλά τα αποτελέσματα, θετικά, αλλά επιδέχονται βελτιώσεων. Ε, δεν θα μιλήσω για τα αποτελέσματα. Αν έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστως να απαντήσω. Αν έχετε ερωτήσεις για τα νούμερα. Ε, υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση που θα δημοσιευτεί σύντομα σχετικά με τα αποτελέσματα του πρώτου στρατηγικού προγράμματος και βέβαια αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα του πρώτου προγράμματος και αντλήσαμε διδάγματα. Ε, είδαμε δηλαδή τα θετικά, τα λιγότερο θετικά, βγάλαμε διδάγματα, τα οποία επίσης αντικατοπτρίζονται στο δεύτερο στρατηγικό πρόγραμμα. το, το όραμα του πρώτου προγράμματος 11-14 ήταν να δημιουργήσει ένα δίκτυο ε, για τα σήματα σχέδια υποδείγματα. Υπήρχε ένας ανταγωνισμός ε, ε, αμοιβών μεταξύ των εθνικών γραφείων που είναι υπεύθυνα να χορηγούν εθνικά δικαιώματα και υπήρχε ε, πάντοτε ένας ανταγωνισμός μεταξύ της ΙΟΥΙΠΟ και των εθνικών γραφείων. Η συνύπαρξη δεν λειτουργούσε καλά. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα να έχουμε καλή συνεργασία που να έχει νόημα, ε, δραστηριότητες, σύγκληση ούτως ώστε οι διαδικασίες, οι τα συστήματα να ευθυγραμμίζονται εις ό,τι αφορά τα ε, διάφορα ε, συστήματα, σχέδια, υποδείγματα και νομίζω ότι εδώ κάναμε μεγάλη πρόοδο. Επίσης ε, είδαμε ότι υπήρχε κατεπίγουσα ανάγκη το, το, ε, καταχωρήσεις ε, να τις θέσουμε υπό έλεγχο. Ε, έχουμε πολλές χιλιάδες, 60.000 περίπου σχέδια. Κάθε χρόνο χιλιάδες καταθέσεις γίνονται, πολλές καταργήσεις, ακυρώσεις και πρέπει όλα αυτά να, έπρεπε να τα θέσουμε υπό έλεγχο. Μετά θέλαμε να μειώσουμε το χρόνο που παίρνει μεταξύ ε, κατάθεσης της αίτησης και της ε, έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης. Και νομίζω ότι είχαμε επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης καταφέραμε να εντάξουμε νέες αρμοδιότητες στο γραφείο που προβλέπονται από την νομοθεσία. Ε, ε, έχουμε ήδη δύο οδηγίε ε, εντάξει. Ε, εδώ υπάρχουν και κάποιοι ευρωβουλευτές που ήταν μέλη του παρατηρητηρίου, το οποίο το έχουμε αναδιαμορφώσει επίσης. Δηλαδή συγκεντρώνουμε στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για τη λήψη των αποφάσεων. Επίση έχουμε αρμοδιότητες στον τομέα των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκτός Ένωσης. Έχουμε τρία τώρα, διότι το ένα ε, ε, όχι, άρχισε χθε ε, προγράμματα διανοητικής ε, ιδιοκτησίας στην Κίνα, την Ινδία και τους επόμενους μήνες κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και στην Νότιο Αμερική, στην, στις χώρες της Καραϊβικής και τέλος πολύ σημαντικό και αυτό βέβαια είναι θέμα που μας ανησυχεί και μας απασχολεί, στην Αφρική επίσης θα έχουμε αρμοδιότητες από όλες αυτές τις ε, περιοχές. Έτσι λοιπόν, από δίκτυο εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, θέλουμε να περάσουμε και να γίνουμε ε, δίκτυο διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο ως ένα βαθμό περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ε, διανοητικής ε, ιδιοκτησίας και θα διέπεται από τους χρήστες. Αν θυμάστε το παρατηρητήριο και οι αρμοδιότητές του είναι οριζόντιες δεν αναφέρονται αποκλειστικά στα εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα, αλλά σε όλα τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησίας. Το εμπορικό απόρριτο ε, δεν είναι καθ' αυτό δικαίωμα, αλλά είναι κοντά. Τώρα που έχουμε θέση υπό έλεγχο το, το, το, το θέμα του χρόνου, ποιότητα στα πλαίσια τα σωστά χρονικά, τώρα θέλουμε προβλεψιμότητα αποφάσεων και ποιότητα αποφάσεων. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Σας είπα ότι το 2010-2010 πήραμε εμπορικά σήματα 90.000 ε, και 60.000 σχέδια και υποδείγματα. Τώρα 130.000 εμπορικά σήματα και 90.000 σχέδια υποδείγματα. Οπότε έχουμε αύξηση 30-40% μέσα σε 4 χρόνια μόνο. Αν έχουμε 130.000 αποφάσεις να πάρουμε από τη μια και 90.000 από την άλλη, πρέπει να αυξήσουμε την συνέπεια των αποφάσεων. Αλλιώς η προβλεψιμότητα των αποφάσεων μειώνεται και το κόστος για τη βιομηχανία αυξάνεται, διότι δεν έχουν προβλέψιμο σύστημα και πρέπει να επενδύσουν πολύ περισσότερα στις νομικές συμβουλές, στους δικηγόρους, ούτως ώστε να φτάσουν στην απόφαση που θεωρούσαν λογική. Θέλουμε λοιπόν να επενδύσουμε περισσότερο στην ποιότητα των ε, εργασιών μας. Ε, ποιότητα και συνέπεια μας ε, ενδιαφέρουν εδώ και κάνουμε προσπάθειες για να έχουμε οδηγίες του γραφείου. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Είναι οδηγίες προς τους νομοθέτες και θέλουμε να το διευρύνουμε αυτό για να καλύψουμε, θα έλεγα, και το σύστημα IPC ολόκληρο. Την ερμηνεία που δίνουμε στην νομοθεσία και την ερμηνεία που δίνουν τα κράτη-μέλη. Γιατί βλέπουμε ότι κατά το παρελθόν τα θεσμικά όργανα έκαναν προσπάθεια ε, προς την κατεύθυνση νομικής σύγκλησης μεταξύ των συστημάτων. Όταν όμως μεταφέρεται η νομοθεσία στα κράτη-μέλη της Ένωσης, τι συμφέρει, παρατηρείται απόκληση. Η απόκληση δηλαδή παραμένει ή και αυξάνεται. Γιατί όταν μιλάμε για τον μέσο καταναλωτή, αγαπητέ μου πρόεδρε, ή την πιθανότητα σύγχυσης μέσο καταναλωτή, όταν μιλάμε για ομοιότητα μεταξύ ε, προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών, αυτό πώς θα μεταφραστεί στον νόμο. Δεν γίνεται. Η, μεταφορά, η τέχνη μεταφοράς δηλαδή στην, ε, στο εσωτερικό δίκαιο, η πράξη της μεταφοράς ε, που ερμηνεύει, ε, ε, στηρίζεται σε ερμηνεία οδηγιών και αυτό αυξάνει την απόκληση. Τα επόμενα χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητεί για την κατεξουσιοδότηση, τις εκτελεστικές πράξεις και τα κράτη-μέλη θα συζητούν για την μεταφορά της οδηγίας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα είμαστε ευθυγραμμισμένοι ως προς την ερμηνεία που δίνουμε στα διάφορα στοιχεία με βάση το έργο και του Κοινοβουλίου. Ε, έτσι θα έχουμε ένα πρόγραμμα σύγκλησης και θα διασφαλίσουμε ότι θα συνεπάρχουν τα συστήματα καλύτερα. Και αν τα καταφέρουμε εδώ, θα έχουμε μειώσει τα, τα αρνητικά εξωτερικά στοιχεία, τα οποία ε, επιβαρύνουν τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις όταν αλληλεπιδρούν με, τη δημόσια, με τις δημόσιες διοικήσεις. Ε, έχουμε και εξωτερικούς συνεργάτες ε, που εργάζονται στους τομείς ε, σύγκλησης. Δουλεύουμε ομαδικά, πιστεύουμε στην δύναμη των δικτύων. Έχουμε δημιουργήσει δεκάδες εσωτερικά δίκτυα τα οποία φέρνουν γνώση σε ό,τι κάνουμε, αποτελεσματικότητα επίσης. Έχουμε μεταφέρει αυτή την άποψη για τα δίκτυα και προς το εξωτερικό και το γραφείο ασχολείται και στηρίζεται σε ε, δίκτυα με ε, τους εθνικούς οργανισμούς, επίσης ε, και το, δίκτυο, ε, το παρατηρητήριο κατ' ουσίαν είναι δίκτυο και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στα δίκτυα γιατί δεν μπορούμε να δρούμε απομονωμένα πλέον. Και θα είμαστε πολύ πιο ισχυροί αν μοιραζόμαστε την γνώση και φροντίσουμε όλες οι συνιστώσεις να λαμβάνονται υπόψη στην εξίσωση πριν αποφασίσουμε ε, για κάποιο βήμα που θα κάνουμε στο μέλλον και πώς θα κινηθούμε. Τέλος, πιστεύουμε ότι σε πέντε χρόνια από τώρα θα έχουμε φέρει μια κουλτούρα μέσα στο γραφείο ώστε πέρα από την καλύτερη αξιολόγηση του κόστους δραστηριοτήτων με βάση τον προϋπολογισμό βάση δραστηριοτήτων ή των έργων για τη διαχείριση του προγράμματος, θα έχουμε φέρει μια κουλτούρα που θα έχει επιφέρει αλλαγές. Πριν υπολογίζαμε κυρίως τα ωφέλη από τα έργα. Τώρα θέλουμε να ε, τα ωφέλη από οτιδήποτε κάνουμε. Ποιότητα ε, υπηρεσιών για τους χρήστες, ποιότητα σε ό,τι αφορά ε, ε, ωφέλη σε ό,τι αφορά ε, την μείωση των ισοδυνάμων πλήρους χρόνου, ε, ωφέλη σε ό,τι αφορά την αξία στην αγορά. Επικεντρωνόμαστε στα ωφέλη παντού και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δείξουμε στα τρία θεσμικά όργανα πώς χρησιμοποιούμε τους πόρους μας και ποια είναι τα ωφέλη που έχουμε εκτιμήσει ότι θα έχουμε και τα ωφέλη που θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ε, πάνω, ε, μετά από τις επενδύσεις που θα κάνουμε. Ε, τώρα έχουμε ένα πιο αφοσιωμένο γραφείο και προσωπικό. Ακόμα είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να λύσουμε. Πρέπει να ανοιχτούμε περισσότερο. Όσο περισσότερο συνεργάζεται το προσωπικό, τόσο καλύτερα θα είναι οι υπηρεσίες, τόσο καλύτερα θα είναι τα προγράμματα και τα έργα. Θα πρέπει να ανακαινήσουμε τα συστήματά μας σε μηχανοργάνωσης. Είναι δαπανηρό αυτό, αλλά θα πρέπει να το ανακαινήσουμε. Αξίζει, όπως και το τμήμα ανθρωπίνων πόρων και τα επιχειρησιακά μας συστήματα, ούτως ώστε να έχουμε αποτελεσματικότητα καλύτερη στο γραφείο και έτσι θα βοηθήσουμε και τη βιομηχανία και θα ε, αυξηθεί και εκεί η αποτελεσματικότητα. Ε, ορισμένα στοιχεία ε, σας τα παρουσίασα μέσα σε ένα τέταρτο περίπου ε, στοιχεία του στρατηγικού προγράμματος και προτιμώ για όσα δεν είπα να απαντήσω σε ερωτήσεις και έτσι να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίαση του πολιετούς αυτού στρατηγικού προγράμματος, το οποίο αναμφίβολα είναι φιλόδοξο. Και είμαι απολύτως σίγουρος ότι είναι φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό συνάμα δεδομένων των επιτυχιών που έχει σημειώσει το γραφείο υπό τη δική σας διεύθυνση, υπό τη δική σας καθοδήγηση. Δημιούργησε το μοναδικό πρόβλημα του δημοσιονομικού πλεονάσματος και ελπίζω να βοηθήσαμε να αντιμετωπιστεί αυτό. Πράγματι, απαντάει ο μιλητής. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο, η κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Πρόεδρο Καμπίνο για την παρουσίασή του. Βρίσκω πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το πολυετήσιο στρατηγικό σας σχέδιο δίδει τόση σημασία στη βελτίωση των βάσεων δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων για το IP είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τονίζουμε και να υπογραμμίζουμε συνεχώς. Θα είναι σε θέση οι βάσεις δεδομένων αυτές να μας επιλύσουν προβλήματα σε σχέση με τα δικαιώματα ε, στο διαδίκτυο. Πόσο, μέχρι πού θα φτάσετε ε, ως αυτό. Η Επιτροπή μας έχει δουλέψει πολύ για τις, ε, στο θέμα των βάσεων δεδομένων και των ε, αρχείων ε, εκτός διαδικτύου. Το Offenworks. Works. Μπορεί κανείς να πλοηγηθεί εκεί. Όμως ο κάτοχος του δικαιώματος μπορεί για τα ορφανά έργα, ε, είναι πιο εύκολο ο κάτοχος να το διεκδικήσει, αλλά ενδεχομένως εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ένα ορφανό έργο, μπορεί να αποσύρει, να ε, συγκεντρώσει όλες αυτές τις πληροφορίες και να το χρησιμοποιήσει με αρκετή νομική ασφάλεια γιατί υπάρχουν και αυτά και θα έπρεπε η χρήση τους να είναι πιο εύκολη. Αναφέρεστε στα εμπορικά μυστικά και στις βάσεις δεδομένων. Είπατε ότι το εμπορικό απόρριτο δεν είναι δικαίωμα IP και θα πρέπει αυτό να το τονίζουμε. Στην οδηγία για τις ε, βάσης δεδομένων η οποία θα ψηφιστεί τον Απρίλιο στην Ολομέλεια δεν προβλέπεται ε, παρέκκληση και εξαίρεση. Ποια είναι η απόψή σας γι' αυτό. Και Δύσκολο είναι να έχουμε μια βάση δεδομένων για εμπορικά απόρριτα, τα οποία είναι απόρριτα και μυστικά εξορισμού. Δύσκολο να το διανοηθώ πώς, ποια μορφή θα έχει, τι θα περιλαμβάνει. Έχουμε και τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά και έχουμε υποστεί κριτική για την υφιστάμενη βάση δεδομένων και το sui generis αυτό δικαίωμα. Και ένας τρόπος να λυθούν αυτά τα προβλήματα, και το έχουμε συζητήσει και με την Προεδρία του Συμβουλίου και με την Επιτροπή, είναι το εξής να έχουμε ε, εγγραφή για το δικαιώματα σου ή και και νομίζω ότι το IPO θα ε, καλωσόριζε μια τέτοια εξέλιξη. Και κάτι που δεν αποτελεί μέρος του πολιετούς προγράμματός σας. Όμως, αφού πρόσφατα συνεδρίασε η ομάδα εργασίας για το ε, παρατηρητήριο και συζητήθηκε το θέμα της συμμετοχής της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στο παρατηρητήριο. Πώς θα το βελτιώσετε αυτό. Και τέλος, ε, θέλω να σχολιάσω μια απόφαση συγκεκριμένη που έλαβε το Συμβούλιο ε, του IPO για τα trademark, για τα εμπορικά σήματα. Ότι δηλαδή δόθηκε ένα εμπορικό σήμα για το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Και ποιο είναι το θέμα, ότι αρχικά ο υπάλληλο είχε απορρίψει αυτή τη διεκδίκηση. Είχε πει ότι είναι μέλο τη κληρονομιά μα, είναι μέρο τη ιστορία μα το ημερολόγιο τη Άννας Φρανκ. Και δεν θα πρέπει η ιστορία να είναι ανοιχτή στην εμπορική εκμετάλλευση μέσω του εμπορικού σήματος. Και μετά απορρίφθηκε η απόφαση αυτή και είπε κανείς ότι αφού κανείς μπορεί να κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα Χάρι Πότερ, γιατί δεν μπορεί να κατοχυρώσει και το εμπορικό σήμα της Άννας Φραγκ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και κάποια στιγμή η ιστορία θα πρέπει να ανήκει στη δημόσια σφαίρα, να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε ε, ελεύθερα χωρίς δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας, IP δηλαδή. Πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσετε αυτά, πώς θα τα αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Δεν θα έλεγα ότι τα εμπορικά απόρριτα δεν ανήκουν στην πνευματική διανοητική ιδιοκτησία. Δεν θα πήγαινα τόσο μακριά, γιατί τα εμπορικά απόρριτα βασίζονται στη τεχνογνωσία και στο TRIPS ε, θεωρείται η τεχνογνωσία ότι είναι μέρος της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα ήθελα δύο πράγματα να πω μόνο. Πρώτον, ότι Το γραφείο λειτουργεί υποδειγματικά με τα εργαλεία που διαθέτει. Αυτή την εντύπωση έχω και βλέπω ότι με την πάροδο των ετών υπάρχει ένα εργαλείο ελέγχου εξαιρετικά αποτελεσματικό. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Μπορούμε να πλοηγηθούμε, να συμβουληθούμε σε αυτές τις βάσεις δεδομένων. Το γραφείο λοιπόν ε, ε, διοικείται πάρα πολύ σωστά και καλά και το λέω αυτό δημόσια και δεν είναι σύνηθες αυτό σε άλλες υπηρεσίες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εξουσιοδοτεί δεν είχαμε τόσο καλά αποτελέσματα και θέλω λοιπόν δημόσια να πω ότι το γραφείο σας λειτουργεί ε, υποδειγματικά και σας συγχαίρω. Ωστόσο, Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ήμουνα σε μια άλλη συνεδρίαση και η παρουσία μου εκεί ήταν απαραίτητη. Με ανησυχεί ιδιαίτερως η λειτουργία του παρατηρητηρίου και εκεί θα πρέπει να τεθεί επικεφαλής κάποιος εξίσου αξιόλογος όσο και εσείς Εγώ είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού, υπέρ της αλλαγής στην Ευρώπη Είμαι υπέρ της ενίσχυσης της ψηφιακής πολιτικής, η οποία θα πρέπει να διαχειριστεί περισσότερο στη χώρα μας, χωρίς όμως να ε, καταρριφθούν όλα τα δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής διδιοκτησίας, δικαιώματα που αποτελούν τον ε, εντός εισαγωγικών ορυκτό πλούτο, ε, πάνω, ε, στον οποίο δημιουργείται και παράγεται τελικά πολύ περισσότερο έργο. Ευχαριστώ, κύριο Τζαμπά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω ερωτήσεις να απευθύνω στον επικεφαλής του γραφείου. Θα ήθελα, κύριε Καμπίνος, να σας συγχαρώ για τα στοιχεία, για τις πληροφορίες, τα οποία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ελπίζω να συνεργαστείτε καλά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Κάνετε πράγματα πολύ χρήσιμα και πρέπει να συνεχίσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια. Καλοδεχούμενα, αλλά θα συνεχίσουμε εμείς να χαμογελάμε ελπίζω για την Κυρία Ρέντα, πολύ καλές ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις είναι εντός της στρατηγικού μας σχεδίου, κάποιες άλλες είναι εκτός στρατηγικού σχεδίου. Έχουμε εδώ και τον διευθυντή του παρατηρητηρίου που μπορεί να συμπληρώσει τις απαντήσεις μου. Έχουμε επίσης και από άλλες υπηρεσίες της οργάνωσής μας υπευθύνου και αν ο πρόεδρος το επιτρέψει ίσως να θελήσουν να συμπληρώσουν τις παρατήρησεις μου. Έχετε δίκιο στην πρώτη σας παρατήρηση κύριε Πρέντα, Ρέντα. Ε, ξέρω ότι τα θέματα τα οποία θίξατε είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει θέμα καταγραφής για τέτοιου είδους ε, σήματα. Αλλά ένα τέτοιο ε, εμπορικό σήμα βέβαια, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό σχέδιο, ε, τα πρότυπα μπορούν να καταγραφούν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αν είναι υποχρεωτικό ή μη υποχρεωτικό να καταγραφούν είναι αλήθεια ότι θα πρέπει η δημόσια υπηρεσία να καταστήσει την πληροφορία διαθέσιμη στην κοινωνία γενικότερα έτσι ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και η υπόλοιπη κοινωνία να αμφισβητήσει ίσως τέτοιου είδους δικαιώματα ή να αναγνωρίσει την ύπαρξη ενός τέτοιου αποκλειστικού δικαιώματος. Το είδαμε αυτό σε πάρα πολλές ε, περιοχές, στον τομέα της ταξινόμησης, στον τομέα της επιβολής. Έχουμε δημιουργήσει τεράστιες τράπεζες δεδομένων με 40 εκατομμύρια εμπορικά σήματα τα οποία μπορούν να αναζητηθούν δωρεάν από 50 χώρες. Από ό,τι ακούω και το Ισραήλ θέλει να πάρει μέρος σε αυτήν την ε, τη βάση δεδομένων, το ίδιο και η Κίνα. Ε, κυρία Ρέντα, αν θέλετε να προστατεύσετε το σήμα σας στην Κίνα ε, σήμερα, πώς το κάνετε. Πρέπει να πάτε στην Κίνα, στην αρμόδια υπηρεσία και να δαπανίσετε χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα τώρα πια να καταστήσουμε την επιβολή ε, δεδομένη ενός συγκεκριμένου εμπορικού σύστηματος. Αυτό αφορά και την Κίνα, αφορά και την Ιαπωνία και ιδιαίτερα στα σχέδια έχουμε μια τράπεζα δεδομένων με 10 εκατομμύρια σχέδια την οποία μπορείτε να αναζητήσετε δωρεάν. Απαιτείται όμως να αυξηθούν ακόμα περισσότερο αυτές οι βάσεις δεδομένων και να βελτιωθούν σε επίπεδο ευκολίας χρήσης πρόσφατα, νομίζω και για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Έχουν και αντίστοιχα προγράμματα στην Κορέα και στην Κίνα, αλλά τα δικά μας είναι καλύτερα γιατί είναι ευρωπαϊκά. Έχουν ε, ένα μέσο αναζήτησης εμπορικών ε, σημάτων σε εικόνες, όχι κείμενας, εικόνες. Και αν τώρα τα επόμενα πέντε χρόνια μπορώ να καταστήσω δωρεάν στην βιομηχανία μας την έρευνα εικόνων για σχέδια δηλαδή αποκλειστικά είναι κάτι το βασικό γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καινοτομική δραστηριότητα. Οποιοδήποτε σχέδιο έχει καταχωρηθεί είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε άμεση πρόσβαση. Δεν ξέρουμε ακριβώς ε, ποια είναι τα σχέδια που προστατεύονται και σε ποιες περιοχές του κόσμου. Έχουμε βέβαια τη συλλογή των Κινέζων σε σχέση με τα εμπορικά σχέδια. Υπάρχει μια τέτοια διαδικασία στην Κίνα και στο τέλος του χρόνου θα είναι διαθέσιμη και σε μας. Θα το μελετήσουμε το θέμα αυτό λοιπόν. Να προσπαθήσουμε να δούμε πώς κάποιος ο οποίος δημιουργεί κάτι στην Ευρώπη, είτε αυτό είναι είδος τροφίμων που καλύπτεται από μία συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίες ή κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε άλλο πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες δυνατότητες προστασίας και να αποδείξει στα δικαστήρια αν το χρειαστεί ότι έχει δημιουργήσει κάτι και έχει καταχωρήσει την δημιουργία του σε μια δεδομένη βάση είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε σε ευρωπαϊκό, έχουμε σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο, έχουμε σε επίπεδο εθνικό σε ορισμένες χώρες, στον Πενελούξ επίσης. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξουν νομοθετικές αλλαγές. Δεν είμαι πάντα υπέρ αυτών των νομοθετικών αλλαγών, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν μερικές φορές εύκολες λύσεις που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών με ένα ή πέντε ευρώ μπορεί κανείς ή και δωρεάν ακόμα να ενημερώνεται. Εσείς θα μπορείτε στο όνομά σας να καταθέτετε την πρότασή σας, να αποθηκεύετε σε μία τράπεζα δεδομένων, να λέτε ότι εσείς δημιουργήσατε το συγκεκριμένο αυτό στοιχείο και ε, η κυρία Ρέντα αν της αμφισβητηθεί το δικαίωμα αυτό την παραπέμπουν στο δικαστήριο και στο δικαστήριο θα πει ότι κοιτάξτε εγώ κατοχύρωσα το δημιούργημά μου συνεπώς η δίωξη εις βάρος μου είναι ατεκμηρίωτη. Λοιπόν, ε, χωρίς την ανάγκη να καταφεύγει κανείς σε συμβολιογράφος γιατί σήμερα είναι η μοναδική λύση η οποία υπάρχει αλλά αν υπάρχει μια δημόσια δυνατότητα καταγραφής όλων αυτών των σχεδίων και προτύπων, τότε θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις περιπλοκότητες των νόμων, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ε, και νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι απλά θα πρέπει να διευρύνουμε ακόμα τον ρόλο των τραπεζών δεδομένων. Αυτό το οποίο ενθυμούμε είναι ότι σαν κανόνας τώρα και για την συνέχεια της υπηρεσίας μου υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης μιας mission a study in order to draw a baseline against which then this volume of litigation σε σχέση που υπάρχει μια νομική διαφορά υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθηθεί η συνέπεια της εφαρμογής της απόφασης που έχει ληφθεί σε μια δεδομένη φάση. Ε, αυτά κυρία Ρέντα. Τώρα και για τα σου γένερης, ε, δεν υπάρχει γνωμοδότηση συγκεκριμένη από πλευράς μου, δεν έχει νόημα να σας δώσω την προσωπική μου άποψη, αλλά εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο καλούμεθα να κάνουμε. Ε, μεγαλύτερη εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Φυσικά έχετε δίκιο. Εμείς κάναμε μία μελέτη για να κατανοήσουμε το επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών και είναι σαφές πλέον, αν και πήραμε πάνω από 80% θετικές απαντήσεις, είναι σαφές ότι θα πρέπει εμείς να επανεξετάσουμε ε, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών γιατί οι 50% είναι ικανοποιημένες και οι υπόλοιποι 50% όχι ε, ιδιαίτερα ικανοποιημένες. Θα συνεχίσουμε αλλά ελπίζω να σας έπεισα λίγο σήμερα ότι προσπαθούμε εμείς να λάβουμε υπόψη μας όλες τις απόψεις και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Θυμάμαι σε μία συνάντηση με εκπροσώπους ομάδων χριστών που είπατε α, εσείς είστε ο, βιομη... ο δικηγόρος της βιομηχανίας, ο συνήγορος της βιομηχανίας. Λέω όχι, εγώ δεν είναι ο ρόλος μου. Εγώ έχω τον ρόλο τον οποίο μου έχει δώσει ο νομοθέτης τον κανονισμό και αυτό προσπαθώ να φέρω εις πέρας. Δεν υπερασπίζομαι εγώ την προστασία συγκεκριμένων συμφερόντων, είμαι εδώ για να ακούσω όλους τους εμπλεκομένους και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας επί τη βάση αυτής της μεθοδολογίας που θεωρούμε αξιόλογη και η οποία μπορεί πάντα να βελτιωθεί και επί τη βάση επίσης δεδομένων συγκεκριμένων των οποίων η συλλογή και αυτή μπορεί να βελτιωθεί και με όλα αυτά παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Συνεπώς δεν θέλουμε εμείς ε, να προχωρήσουμε ε, σε, βιαστικά, σε βιαστικές αποφάσεις, το έχουμε πει αυτό και θα συνεχίσουμε να είμαστε δεκτικοί και ελπίζω εκεί να μας βοηθήσετε. Εμείς δείξαμε ότι μπορούμε με τις επιμέρους αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση του κοινού στις τράπεζες δεδομένων δείχνουμε εν πάση περιπτώσει ότι κάνουμε περισσότερα ίσως από όσα χρειάστηκαν και στην ουσία αυτό που μας ζητήθηκε είναι να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες τράπεζες δεδομένων και αυτό το οποίο ε, προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Ε, και να το κάνουμε βέβαια χρήσιμο, εύχριστο ταυτόχρονα δεν έχει νόημα να τα φτιάχνουμε αυτά και να τα εγκαταλείπουμε μετά. Πιέζουν να εφαρμόσουν τις ε, συγκεκριμένες οδηγίες. Δημιουργούμε επίσης ε, περαιτέρω βάσεις δεδομένων. έτσι ώστε αυτές οι τράπεζες δεδομένων να είναι πλούσιες και εύχριστες. Είναι βασικό για μας αυτή η προσπάθεια και τα θέματα, τα, τα μέσα πληροφορικής που χρησιμοποιούμε είναι ένα μέσο, δεν είναι αυτός σκοπός και προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κυρία Ρέντα, κάθε φορά που τα τελευταία χρόνια of... independent. In fact, το θέμα της ανεξαρτησίας. Οι ομάδες κρίσεων ε, είναι ανεξάρτητες, δεν δέχονται οδηγίες ε, από κανέναν και ούτε φυσικά από, από εμένα, που έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ιδιαίτερα ικανός σε αυτά, και είναι ε, ομάδες οι οποίες παίρνουν τις αποφάσεις τους εντελώς αυτόνομα. Εμείς έχουμε μετατρέψει τον κανονισμό για τα εμπορικά σήματα σε, σε... σε επίπεδο ε, καθοδηγητικών γραμμών. Προσπαθούμε εμείς να επιτρέψουμε την ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών, να ερχόμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις ομάδες των πολιτών, να συλλέγουμε όλα τα στοιχεία Ε, οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές δεν είναι δεσμευτικές βέβαια, αλλά παρόλα αυτά και ε, σε σχέση με τις αποφάσεις των δικαστηρίων μιλάμε για ένα έγγραφο αναφοράς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει τυφλά να σεβαστούμε, αλλά σίγουρα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και θα πρέπει να πείσουμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι είναι καλό να υπάρχει μια συγκλίνουσα ερμηνεία του νόμου, αλλά δεν μπορώ να υποχρεώσω και έτσι και αλλιώ ε, το σε επίπεδο εφετείας αν θέλετε η αρμόδια υπηρεσία είναι αυτή η οποία παίρνει τις ε, ε, ανεξάρτητες αποφάσεις. Η προσωπική μου άποψη δεν έχει σημασία, μπορούμε αν θέλετε ε, να συμφάγουμε και να συζητήσουμε και τις προσωπικές μου απόψεις για όλα αυτά. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στις ερωτήσεις σας, σας ευχαριστώ πολύ και αν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Καμπίνιος για τις εξηγήσει σας και τις απαντήσεις σας. Δεν ξέρω αν κανένα συνάδελφος uh, θέλει κάτι τώρα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι εδώ και σας ευχαριστώ που με τόσο πάθος παρουσιάσατε την υπόθεσή σας. Ευχαριστούμε.